propose d'ouvrir notre euh, séance de travail. Euh, l'ordre du jour vous. Καλημέρα σα. Έχετε την ημερήσια διάταξη, δεν έχουν ε, προταθεί αλλαγέ, οπότε αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει υιοθετείτε. Και όσον αφορά τι ανακοινώσει, δεν έχω τίποτα ιδιαίτερο. Οπότε αυτό που σα προτείνω είναι να περάσουμε αμέσω στο σημείο 3 και να δώσουμε το λόγο στην κυρία Ρεζίνα Μπάστος. Για αυτή την υπόθεση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής όσον αφορά την απλοποίηση ορισμένων απαιτήσεων και τη δημοσιονομική διαχείριση. Θα θυμάστε πως πρόκειται για ένα παλιό θέμα κατά κάποιο τρόπο γιατί συνδέεται με αυτό που, που, που αποκαλείται πλάνο ανάκαμψης ε, από το 2008 το έχουμε συζητήσει ένα πακέτο μέτρων δηλαδή μια δέσμη μέτρων και ότι Μέχρι στιγμής είναι μπλοκαρισμένο αυτό το θέμα γιατί επειδή δεν έγινε σύμφωνα με τη διαδικασία η εμπλοκή του Κοινοβουλίου, το αίτημά μας για ενισχυμένη συνεργασία ελήφθη υπόψη πολύ αργά, ενώ η αρμόδια από τις ουσίες Επιτροπή, δηλαδή η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων, είχε η ίδια ε, προτρέξει των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Είμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν κάπως κρίσιμη. Ακόμα και αν η υπεύθυνη επί της ουσίας Επιτροπή ακόμα είναι υποδιαπραγμάτευση με το Συμβούλιο με, πριν από τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο και μέσω μιας καταχραστικής ερμηνείας του κανονισμού, όπως έχω εγώ την εντύπωση, μας ζήτησαν να κάνουμε μια γνωμοδότηση σε ενισχυμένη ε, συνεργασία και νομίζω εγώ ωστόσο πως είναι σκόπιμο η Επιτροπή μας να μπορέσει να φέρει γνώμη σε αυτό το θέμα. Γιατί το κοινωνικό ταμείο που είναι σημαντικό όσον αφορά το κονδύλι και ε, επειδή πρόκειται για σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να γνωμοδοτήσουμε να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί δέχτηκε κάπως να τα στριμώξει στο χρονοδιάγραμμά της και μπορέσαμε να φτιάξουμε κάτι που στέκει με βάση το χρονοδιάγραμμα της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής. Έχετε το λόγο κυρία εισηγήτρια. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποια είναι η διαδικασία εντός της οποίας παρεμβαίνετε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για το ιστορικό που μας δώσατε, για την συγκεκριμένη έκθεση, μάλλον γνωμοδότηση. Να σας δώσω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για το ποια ακριβώς ήταν η δουλειά μου σε σχέση με την πρόταση μεταρρύθμισης των τριών ταμείων, του Κοινωνικού Ταμείου, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής. Όπως γνωρίζετε, διανύουμε μια χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση εξαιρετικά σοβαρή, πράγμα το οποίο πιέζει τους εθνικούς πόρους. Είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για να βληθούν οι πίεση αυτή να μπορέσουμε έτσι να φτάσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο σε πιο αποδοτικό και ταχύ τρόπο χρήσης των κοινοτικών πόρων καθώς Πιστεύουμε πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουν να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη και οι δικαιούχοι, δηλαδή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Γνωρίζουμε πως η πραγματική οικονομία βασίζεται βασικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ότι η κοινοτική πόρη αυτών των προγραμμάτων συνοχής μπορεί να αποτελέσει έναν βασικό θεμέλιο για να τεθούν οι βάσεις για μια νέα ανάκαμψη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο κινητήρας της, οικον... ευρωπαϊκής οικονομίας και οι βασικοί φορείς τη βιώσιμη ανάπτυξης φτιάχνουν θέσεις απασχόλησης σε ποσότητα και ποιότητα. Φτάνει να δει κανεί, ότι 25 εκατομμύρια μικρομεσαίε αποτελούν έναν αριθμό που υπάρχει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιπροσωπεύει το 90% των επιχειρήσεων τη Ένωση. και πρόκειται για 25 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Οι προσπάθειες λοιπόν, ξέρουμε μάλλον πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ συχνά πολύ ευάλωτες. Ε, ε, ιδιαίτερα στο, στους τομείς ε, της, ε, ε οικοδομή, της οικοδομής αλλά και της κατασκευής επίπλων. Πρόκειται όμως για το 80% των θέσεων απασχόλησης στους δύο αυτούς τομείς και γι' αυτό και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ιδιαίτερα έδωσαν προσοχή σε αυτό το φαινόμενο της χρήσης και της απλοποίησης της χρήσης των πόρων των τριών ταμείων της πολιτικής συνοχής που χωρίς καμιά αμφιβολία είναι το απαραίτητο όργανο για την εφαρμογή των πολιτικών, την υποβοήθηση μάλλον των πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πρόκειται για μέτρα τα οποία καθιστούν ε, την χρήση αυτών των ε, ταμείων, αυτών των κονδυλίων πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική. Ε, Ω προ αυτή την κατένθεση, δούλεψε η αρμόδια επί ε, επιτροπή μέσω του εισηγητή τη κυρίου Κύρι Λόφ και επίσης προς αυτή την κατεύθυνση έχει κατευθυνθεί δικιά μου εργασία σε αυτή τη γνωμοδότηση. Η γνωμοδότησή μου λοιπόν είναι πολύ απλή. Δύο τροπολογίες ε, για διαγραφή έχουν ε, υποβληθεί, όπως και για το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Περιφερειών. Η μία ενισχύει την βελτιστοποιημένη χρήση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστούν τα, ε, τα δραστήρια μέτρα στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται να υπάρξει μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και αύξηση των θέσεων απασχόλησης με μέσα όπως αυτά εδώ, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να επανέλθουν εκ νέου στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, Αφού δώσαμε το ιστορικό και τις διάφορες φάσεις ε, της διαδικαστικής θα πρέπει να σας πω ότι η ημερομηνία για την υποβολή ε, τροπολογιών έχει προσαρμοστεί στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει επιταχυνθεί ώστε η έκθεση αυτή να μπορέσει να εγκριθεί εντός κάποιου λογικού χρονικού διαστήματος ώστε να έχουμε την ε, αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε και όσον αφορά την εφαρμογή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σρότερ και μετά κυρία Λίν. Όλες οι αντιπρόεδροι εδώ έχουν κινητοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την εισηγήτρια, για τα όσα μας εξέθεσε, αλλά διαφωνώ μαζί της. Δεν με την άποψή της. Έχουμε μια τροποποίηση εδώ του κανονισμού των Ευρωπαϊκών Διαθετικών Ταμείων και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα εξή τρία κεντρικά ζητήματα. Το πρώτο αφορά τη δική μας Επιτροπή ουσιαστικά και την αρμοδιότητά του και κατά την άποψή μου ήταν και ο βασικός λόγος για τον οποίο η Πρόεδρος αγωνίστηκε να έχουμε καλύτερη θέση ε, το όλο εγχείρημα ως Επιτροπή. Και ποιο λοιπόν είναι το ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα χρηματοδοτείται για κάποιο διάστημα 100% για να μην έχουν συγχρηματοδότηση τα κράτη-μέλη για να μπορούν να τρέξουν σε πόρους του κονδυλίου του ταμείου αυτού. Αυτό το απέρριψε το Συμβούλιο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Και φταίει και ο κύριος Κύριλοφ γι' αυτό. Το Κοινοβούλιο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε θέση πριν από το Συμβούλιο. Δηλαδή ο κύριος Κύριλοφ υιοθέτησε ουσιαστικά τη θέση ε, του Συμβουλίου με καμιά δυο προσθήκες και τίθεται το ερώτημα εάν ε, θα συμφωνήσει η Επιτροπή μας ή αν θα προσπαθήσει και πάλι να ξαναδεί αυτό το θέμα της 100% χρηματοδότησης, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Δεν είναι περισσότερα χρήματα, προσέξτε. Ε, ε, απλώς είναι να προωθηθούν κάποια προγράμματα, κάποια έργα εκεί που έχουν αποτελματωθεί λόγω της έλλειψης ή χρηματοδότησης. Και τα χρήματα λοιπόν παραμένουν αυτά στη διάθεση των κρατών μελών. Και αργότερα όταν βελτιωθούν τα πράγματα τότε ε, θα δοθεί η κρατική συγχρηματοδότηση. Πρόκειται για προκαταβολές. Δεν, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς έχουμε καθυστέρηση στην απορρόφηση. Είναι βασικό αυτό το θέμα και το Συμβούλιο το απέρριψε. Θέλουμε να συγκρουστούμε με το Συμβούλιο. Θέλουμε ε, επενδύσεις και θέσεις απασχόλησης. Τότε αυτή θα ήταν η σωστή θέση να το κάνουμε και να το δηλώσουμε. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, δεν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι τεράστια έργα. Τεράστια έργα πάνω από 25 εκατομμύρια μέχρι 50 εκατομμύρια σε αυτή την τάξη μεγέθους είναι. Αν θα πρέπει να τα εγκρίνει η Κομισιόν ή όχι. Όταν είναι μια τάξη μεταξύ 25 και 50 εκατομμυρίων. Εγώ συμφωνώ να τα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να έχουμε και ένα δεύτερο έλεγχο, να μην έχουμε προβλήματα στη διαδικασία και να συμφωνούμε για τα κεντρικά αυτά τα μεγάλα έργα. Και αν δεν συμβαίνει αυτό είναι πρόβλημα. Και ένα τρίτο, επίση πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή και είναι ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη ελάφρυνση, διευκόλυνση με την κατάσταση των επιχειρήσεων. Δηλαδή θα ε, εισπράττει κανείς τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τα διορθωτικά ταμεία και θα παίρνει την ε, επιχείρησή του και θα φεύγει. Όχι, θα πρέπει να πούμε όποιος παίρνει ενίσχυση από τα διορθωτικά ταμεία θα πρέπει να παραμένει επί τόπου και ε, τις επιδοτήσεις αυτές να τις... Ε, επενδύει για δημιουργία θέσεων απασχόληση. Δεν θα πρέπει γενικά να ευλογούμε αυτά που αποφασίζει το Συμβούλιο, να έχουμε δικιά μα θέση, έτσι κι εμεί εμείς τροπολογίες θα κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ η κυρία Λίν και μετά η κυρία Σίπερ. Uh, Έχω κάποιες ανησυχίες για την τροπολογία 2 και τη 4, γιατί αφαίρουν τη δυνατότητα της χρηματοδότησης κατά 100%. Λέει στο αρχικό κείμενο ότι είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί για κάποια περιορισμένη χρονική περίοδο. Αυτό είναι όλο. Δεν λέει εσάι γιατί υπάρχουν συγκεκριμένε ε, και περιορισμοί από τους οποίους εργάζονται τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή. 100% χρηματοδότηση για όσο είναι απαραίτητο, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι κάποια χρήματα του, ταμείου, του κοινωνικού ταμείου δεν περνάνε γιατί η δυνατότητα δεν, ε, δεν έχουν τα κράτη-μέλη για να απελευθερώσουν αυτά τα χρήματα. Νομίζω λοιπόν πω θα ήταν σημαντικό να υπάρχει η δυνατότητα το 100% και ίσω θα πρέπει αυτό να το ξανασκεφτούμε, διότι το να διαγράψουμε αυτό που λέτε στις τροπολογίες 2 και 4 δεν είναι σωστό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πολύ. Το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο ουσιαστικό, είναι και χρονικό. Συμφωνώ με την, πρόοδο, με Πρόεδρο ότι ακριβώς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και καλό θα ήταν η δική μας Επιτροπή να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Εντάξει, μας λυπεί αυτό και είναι πολύ ενοχλητικό. Το θέμα της χρηματοδότησης κατά 100% να σας πω ότι πρώτη φορά που είδα την πρόταση αυτή πέρυσι, σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα για να αντιδράσουμε στην κρίση γρήγορα και να βοηθήσουμε τι περιφέρειες που πλήγονται, όχι τα κράτη. Και θέλω να γίνει αυτή η διάκριση, παρακαλώ. Ε, τι περιφέρειες που πλήττονται, για να έχουν γρήγορα τα χρήματα στη διάθεσή τους. Δεν θέλω να μπω στην προϊστορία καθόλου. Επί τη ουσία όμως έχουμε το εξή πρόβλημα. Το Συμβούλιο και μάλιστα η μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών διαφώνησε με αυτές τις προκαταβολές με νύχια και με δόντια. Ακόμα και αν το Κοινοβούλιο αποφάσιζε τώρα με μεγάλη πλειοψηφία ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 100% χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο, θα μπαίναμε σε μια διελκυστίδα χρονική με διαπραγματεύσεις για ε, συμβιβασμούς και μέχρι το καλοκαίρι δεν θα καταφέρναμε τίποτα και δεν θα βοηθούσαμε κανέναν. Αυτό όμως που θεωρώ σημαντικό είναι να λάβει θέση επί της αρχής η Επιτροπή μας και να πει ότι θεωρούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλή ή κακή επί της αρχής τουλάχιστον για μελλοντικέ διαδικασίες για τα ταμεία να το χρησιμοποιήσουμε ως δυνατότητα, ως ενδεχόμενο καταπολέμησης κρίσεων για να μην χαθεί εντελώς. Τώρα για τις συγκεκριμένες τροπολογίες εμείς που είμαστε και Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να βάλουμε και άλλα θέματα, στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, α πούμε, ω Επιτροπή Απασχόληση, δεν μα ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε τι οποιασδήποτε θέσει απασχόληση, να είναι καλέ, καλά πληρωμένε, ασφαλεί θέσει απασχόληση, να το ξαναπούμε αυτό ξεκάθαρα. Και εκεί που λέμε ε, να μην χάνει ο κόσμος τη δουλειά του και αν τη χάνει να βρίσκει γρήγορα καινούρια. Και αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει στην Επιτροπή μας, ότι θέλουμε νέες θέσεις απασχόλησης ίσης αξίας και ποιότητας όταν κλείνουν επιχειρήσεις να μην πέφτουν ε, σε ένα κατήφορο οι εργαζόμενοι να ε, να δέχονται θέσεις απασχόλησης επισφαλής με κακή αμοιβή. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, συμφωνούμε με το 100% που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώ ορίζουμε την πρόταση και αν μη τι άλλο για το μέλλον να το ξανασκεφτούμε, να μην το απορρίψουμε και να έχουμε μεγαλύτερο βάρος στις τροπολογίες λέγοντας ότι χρειαζόμαστε καλές θέσει απασχόλησης ποιοτικέ με προσόντα για αυτές που δημιουργούνται να είναι εισάξιε με εκείνε που χάνονται, όχι όλο και πιο επισφαλής και κακή ποιότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μέσνερ και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι γεγονό ότι έχουν τεράστια προβλήματα στην αγορά εργασία με την κρίση και καλό είναι να σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ μπορεί να βοηθήσει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και πιο γρήγορα και καλύτερα και απλούστερα να διατίθεται τα χρήματα αυτά. Και αυτό το 100% αρχικά μα φαίνεται καλή ιδέα και ακούγεται καλό. Το πρόβλημα είναι όταν δίνει 100% και όχι για περιορισμένο χρόνο, τότε ε, δημιουργεί εξαρτήσει που δεν είναι καλό πράγμα εντάξει, έκτακτες περιστάσεις να βοηθήσουμε την αγορά, την απασχόληση να αυτοβοηθηθεί, αλλά να μην απεμπολίσουμε γενικά τη συγχρηματοδότηση. Δεν το επιθυμεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε τι, τι θέλουμε για το 100% γιατί το Συμβούλιο το απορρίπτει. Και εγώ θέλω να βοηθήσω τον κόσμο και γρήγορα να αποφασίσουμε. Να είναι στοχευμένη όμως η παρέμβασή μας. Έχω και μια άλλη παρατήρηση γιατί είμαι σκιώδη συγγήτρια από την ομάδα μου. Ε, έχουμε μέχρι την Παρασκευή, νομίζω, ευκαιρία να κάνουμε τροπολογίες ε, και αυτό που έχει σημασία είναι η μετεκπαίδευση να προσανατολίζεται στι ανάγκε και τι απαιτήσει τη αγορά, στη συνεννόηση και στενή επαφή με τις ε, εταιρείε, με την οικονομία. Γιατί αυτοί που δημιουργούν τι θέσει, ξέρουν και τι ανάγκε έχουν. Το ξέρω ότι το λέει η έκθεση, αλλά δεν το λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα, γι' αυτό το βάζω ω τροπολογία συμπληρωματική. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το συντομότερο να πάρουμε απόφαση και με τρόπο που να βοηθάει τον κόσμο στοχευμένα ξαναβρει δουλειά και να βγει από την κρίση. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω και εγώ ότι θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να υποστηρίσουμε την αρχή της συγχρηματοδότησης ή όχι. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι δεν στέλνουμε λεφτά στην περιφέρεια, κοινοτικά κονδύλια και είμαστε εντάξει. Όχι. Η συγχρηματοδότηση, η συνυπευθυνότητα έχει και πολιτική σημασία. Να φροντίζουμε οι θεσμοί, ε, οι περιφέρειες που παίρνουν ευρωπαϊκά κονδύλια να καταλαβαίνουν ότι έχουν συμφέρον να τα χρησιμοποιούν σωστά, αποτελεσματικά και ε, γι' αυτό βάζουν και τα ίδια ε, το χέρι στην τσέπη. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο η συγχρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει καθόλου να την εγκαταλείψουμε. Το Συμβούλιο διαφώνησε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ δύσκολο να συμφωνήσει και το Συμβούλιο, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξή. Αν δεν συμφωνήσουμε τώρα για το μέλλον, να μπορούμε να λέμε ότι να παραμείνει στη δική μα επιτροπή, στη δική μα αρμοδιότητα. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν μπορούμε να πούμε ε, θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία όπου συνδέονται οι επιτροπές τουλάχιστον σε ίδιο επίπεδο να συμμετέχουν και οι δύο. Αυτό θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένο. Δεν μπορεί αυτά τα θέματα να τα διαπραγματεύεται μόνο η Περιφερειακή Επιτροπή. Αυτό είναι βασική μας αρμοδιότητα από πάντα η απασχόληση. Τώρα το θέμα των ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, πολύ σωστά το ρύθμισε η Ρεκίνα Μπάστο στην τροπολογία 3 για τους νέους. Αυτή είναι μία διάσταση αλλά αυτό μπορεί να μεταφερθεί και αλλού. Και μπορεί να συμπληρωθεί αν θέλετε. Και μιλάει και υψηλή, για υψηλή ποιότητα μαθητείας για τους νέους. Την επόμενη φορά θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, συμφωνήσουμε, έχουμε λίγε εβδομάδε. Δεν διαφωνούμε ριζικά, γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλε διαφωνίε. Δεν συμβαίνει αυτό. Η Ρεγίνα μπορεί να κάνει ε, συμβιβασμού και να συνεννοηθεί με τι άλλε πολιτικέ ομάδε και την ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Να κάνω κι εγώ κάποιε συμπληρωματικέ παρατηρήσει. Για τη δική μας Επιτροπή δεν πρέπει να υποτιμηθεί το διακύβευμα. Πρέπει να πάρουμε θέση εδώ στην Επιτροπή για δύο λόγους. Όχι, για τρεις λόγους. Πρώτον, το θέμα της αποτελεσματικότητας των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και η δυσκολία κινητοποίησης των κονδύλιων λόγω αυτού του κανόνα χρηματοδότηση σε μια περίοδο κρίσης όπως η σημερινή ήταν ένα επιχείρημα πάρα πολύ σημαντικό, ούτω ώστε η Κομισιόν στην αρχική της πρόταση να προτείνει τη χρηματοδότηση 100%. Το να ξεχάσουμε την ανάλυση της κρίσης και να ξεχάσουμε ότι κάποια εργαλεία του κοινοτικού προϋπολογισμού πρέπει να προσαρμοστούν στην κρίση. Αυτό είναι νομίζω απλή συνενοχή με το Συμβούλιο, που έχει μόνο ένα στόχο τελικά. Τα δημοσιονομικά του κάθε κράτους μέλους. Ξεχνάμε τη λογική του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Και κατά την άποψή μου αυτόν τον τρόπο εμβαθύνουμε τη δυσκολία και δεν λειτουργεί αποτελεσματικά το, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Τη στιγμή που θα κάνουμε τον απολογισμό των διαφορετικών ταμείων θα καταλάβουμε ότι για τα καινουργια κρατη κράτη-μέλη δεν τα εξοπλίσαμε για να αντιμετωπίσουν την κρίση. Και μάλιστα και πριν την έλευση της κρίσης βρισκόταν σε καταστάσεις δύσκολες. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν παλιά στην Πορτογαλία ή στην Ισπανία πρέπει να προβληματιστούμε. Γιατί αυτά τα ταμεία δεν αναπροσαρμόστηκαν στους στόχους και στην πραγματικότητα των νέων κρατών μελών. Τα οποία έχουν και προβλήματα απορρόφησης των κονδύλιων. Τα ξέρουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν θελήσαμε να θέσουμε το δημοσιονομικό ε, ερώτημα κατά τη διεύρυνση. Δεχτήκαμε αυτό που υπήρχε και το αποτέλεσμα είναι ότι οι συγκλήσεις αυτών των οικονομιών δεν έχουν υλοποιηθεί, είναι δύσκολο θέμα και οι οικονομίες αυτές έχουν ε, πληγεί δυσανάλογα από την κρίση. Αν δεν το πούμε αυτό, στην πραγματικότητα παρετούμαστε από την ευρωπαϊκή δημοσιονομική αποτελεσματικότητα. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση με το Συμβούλιο, θα σας μιλήσω ειλικρινά. Οι ευρωβουλευτές που είναι εδώ παρόντες συνέχεια διατυμπανίζουν ότι έχουν εξουσία. Ότι πρέπει να βελτιωθούν και να διορθωθούν οι, προβλημα... οι προσανατολισμοί του Συμβουλίου γιατί δεν είναι σωστοί. Εδώ ορισμένοι κάποιοι έπαιξαν ουσιαστικά και να προκαθορίσουν τη θέση του Κοινοβουλίου πριν γίνει η δημοκρατική διαβούλευση. Και τελικά γονατίζουμε στη θέση του Συμβουλίου. Γονατίζουμε ενώπιον τη θέση του Συμβουλίου και αυτό είναι απαράδεκτο. Τρίτον, καταλαβαίνω τώρα ότι υπάρχει θέμα κατεπήγοντο. Μα αγαπητοί φίλοι, το Κοινοβούλιο έχει δείξει την ε, στάση ε, ευθύνης. Δεν μπορούμε να ξεπετάμε έτσι μέσα 24 ώρες ένα θέμα. Όταν υπάρχει πολιτική συνένεση, ξέρουμε να κινητοποιούμαστε και να ολοκληρώνουμε μια διαπραγμάτευση εγκαίρως. Το Συμβούλιο προαποφάσισε δηλαδή τη θέση του Κοινοβουλίου και εμείς θα πρέπει να γίνουμε συνένοχοι. Αυτό θα κάνουμε. Ε, Ρεγκίνα Μπάστος, στο λέω φιλικά. Αν θέλετε να κάνουμε μια γνωμοδότηση, θα την κάνουμε. Καταλαβαίνω την ε, συνεισφορά τη τροπολογία 3 όπω παρουσιάστηκε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ μεταξύ μα. Αλλά για την τροπολογία 2 και 4 που αποτελούν τη θέση, την καρδιά της θέσης του κυρίου Κυρίλοφ στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή, τότε τι νόημα έχουν να φτιάχνουμε κι εμείς μια γνωμοδότηση, μόνο και μόνο δηλαδή για να γονατίζουμε ενώπιον της θέσης του Κυρίλοφ. Ο τρόπος με τον οποίο θα τοποθετηθούμε σε αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Τόμα Μάν μας λέει θα τα δούμε την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά θα είναι η μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Αν ξεκινήσουμε από αυτήν την ανάλυση και αν με την πρώτη ευκαιρία που μας δίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο κρίση δεν κάνουμε τίποτα και σταυρώνουμε τα χέρια, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα απορροφηθεί από κάτι άλλο. Θα εξαφανιστεί αν πιστεύουμε αυτό που κάνουμε, αν πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό αυτό το ταμείο για να βοηθήσει τον κόσμο, για να δημιουργήσει σε δύσκολες ε, περιφέρειες θέσεις απασχόλησης, Και μην μου λέτε ότι τα κράτη δεν έχουν πρόβλημα σε χρηματοδότηση σε τέτοιες δυσκολίες ε, κρίσης. Εγώ θέλω να βοηθήσω φυσικά την ε, Ισπανική Προεδρία, θέλω να κινητοποιηθούμε γρήγορα, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε μία θέση μέσα σε ένα σωστό πλαίσιο. Σέβομαι τη δουλειά της ε, εισηγητριάς μας. Αλλά σας λέω ειλικρινά δεν συμμερίζομαι την προσέγγισή σας ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της συγχρηματοδότησης. Δεν ξέρω αν άλλοι θέλουν να πάρουν το λόγο, αλλιώς να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να ολοκληρώσουμε και αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, για τη συμβολή τους στον προβληματισμό. Το θέμα είναι πολύ λεπτό και εγώ θα ξεκινούσα λέγοντας πως ε, μέσα στο πλαίσιο αυτής της ε, κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στην οποία ζούμε εγώ με την ιδέα ότι τα κονδύλια της συνοχής είναι ένα ζωτική σημασία ε, μέσο για να βγούμε από την κρίση. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι αυτή είναι η θέση μου όσον αφορά το ρόλο των ε, ταμείων της συνοχής, του Διαρθωτικού Ταμείου και του Κοινωνικού Ταμείου ως ε, μέσων ε, οικονομικών για να βοηθηθούν τα κρατη να βγουν από την κρίση και να μπουν σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Τώρα βέβαια δεν μπορώ ως ε, εισηγήτρια να κλείσω τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα που έχουμε ενώπιον μας και η πραγματικότητα απαιτεί ρεαλισμό. Εάν αυτή τη στιγμή εμείς ε, σταθούμε άκαμπτοι απέναντι στο θέμα της συγχρηματοδότησης θα μπορούσαμε να μην σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, δηλαδή να παραμένουμε σε μια χρήση τέτοιου, αυτών των κονδυλίων με τρόπο ε, γραφειοκρατικό ενώ θέλουμε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, ιδιαίτερα για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφού είναι ο κατεξοχήν τομέας δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι η η συνέχεια που θα δοθεί στη δική μου έκθεση μαζί με τις ε, τροπολογίες και τις τροπολογίες του κυρίου Κυριλόφ στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, αυτό το στόχο έχουν να επιταχυνθεί η δυνατότητα χρήσης των ταμείων συνοχής να μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο απλοποιημένα από τους δικαιούχους που τα χρειάζονται. Τώρα, είπατε, ρωτήσατε τι θα γίνει στο εγγύς μέλλον με τη μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Ταμείου. Θεωρώ πως θα μπορούσε να αυτό να αποτελέσει μια σημαντική ευκαιρία για, την για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα για την Επιτροπή Επασχόληση, ώστε να απαιτήσουμε από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή μια ιδιαίτερη προσοχή να δώσει στην μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, έτσι ώστε στο πλαίσιο το, το ευρύτερο των, των διευθυντικών ταμείων να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και η πολιτική συνοχής ως μια βασική πολιτική που είναι απαραίτητη και αναντικατάστατη για την έξοδο από την κρίση. Όπως είπε ο συνάδελφος ε, Τόμας Μάνα, εγώ δεν είμαι άκαμπτη στις ε, θέσεις μου. Θα λάβω υπόψη τις ε, απόψεις των συναδέλφων που θα υποβάλουν τροπολογίες μέχρι τις 5 του μηνός. Διατηρώ αυτή τη ρεαλιστική θέση και ε, άποψη ε, για αυτή τη φάση, αλλά και τη διεκδικητική θεστάση όσον αφορά την ρόλο της Επιτροπής Απασχόλησης για τη χρήση όλων αυτών των μέσων στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Νομίζω πως αυτός θα είναι ο στόχος, θα υπάρχει συνένεση γι' αυτόν τον ε, στόχο. Βέβαια μετά θα πρέπει να καθορίσουμε ποια θα είναι η πιο αποτελεσματική θέση της Επιτροπής. Όπως μας θύμισε λοιπόν η συγγήτρια, η ημερομηνία κατάθεσης, ε, το, η προθεσμία μάλλον είναι αύριο ε, το μεσημέρι και έπειτα θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στην επόμενή μας συνεδρίαση της Επιτροπής στις 16 Μαρτίου και ε, θα τις ψηφίσουμε την επομένη, δηλαδή στις 17, γιατί η αρμόδια από τις επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει στις 17 και 18 Μαρτίου. Κλείσαμε την εξέταση αυτού του θέματος σας προτείνω να περάσουμε στο σημείο 4 που είναι η εξέταση των τροπολογιών στο σχέδιο γνωμοδότηση του κ. Όλε Κρίστενσεν για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών και για τις πράξεις επανατιτλοποίησης και τον εποπτικό έλεγχο των μισθολογικών πολιτικών. Ευχαριστώ Øh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις τροπολογίες. Ε, θα προσπαθήσω ε, να επιτύχω ευρεία συνένεση για το θέμα αυτό και να το διαβιβάσουμε ως γνωμοδότηση στην Επιτροπή ε, που είναι αρμόδια για το θέμα αυτό, την οικονομική και νομισματική. Στη Δανία υποχρεώθηκαν να κλείσουν πολλές τράπεζες μετά την κρίση. Και το κράτος ε, επιφορτίστηκε με την εγγύηση των καταθέσεων για να μην χάσουν οι άνθρωποι τα χρήματά τους. Στη Βόρεια Γιουτλάνδη, από όπου κατάγομαι, επί παραδείγματι, ε, πτώχευσε μια τράπεζα και αυτό είχε πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες. Ο κόσμος έχασε όλες του τις αποταμιεύσεις. Τα ε, χρήματα ε, που είχε επενδύσει για τη σύνταξή του σε μετοχές χαθήκανε. Και γνωρίζω λοιπόν από τη χώρα μου, όχι μόνο από την περιφέρειά μου και από άλλες περιφέρειες, ε, ότι οι, οι τράπεζες στη Δανία ανέλαβαν πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Γιατί και οι ε, διοικήσει των τραπεζών, τα υψηλά στελέχη, παίρνουν υψηλότερα μπόνους και αμοιβέ ε, όσο αυξάνεται ε, το κέρδος των τραπεζών του. Δηλαδή, οι τράπεζες αναλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Κάτι τέτοιο θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί στο μέλλον και θα φροντίσουμε να μην επαναληφθεί. Η έκθεση θέλει περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη ισορροπία σε όλο το τραπεζικό κλάδο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος αλλαγής πορείας όταν ε, έχουμε μια στρεβλή κατεύθυνση. Γιατί ξέρετε ότι το μέσο αυτό έχει και πολύ μεγάλη ένταση εργασία, πολύ μεγάλη απασχόληση. Επιτρέψτε μου να πω τώρα στι τροπολογίε. Ο Τόμα Μαν έχει κάνει τι τροπολογίε 40, 45 και 53. Είμαι μεν υπέρ, αλλά πρέπει να σας πω ότι στην 53 ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση. Και η κυρία Τσίμερ έχει κάνει τις τροπολογίες 41, 42, 43 και θα πρότεινα εκεί συμβιβαστικές διατυπώσεις. Για δε τα μισολογικά θα πρέπει να πούμε ότι έχουμε πριμ που είναι 300 πλάσιες από τις κανονικές αμοιβέ ε, των ε, στελεχών της τράπεζας, των εργαζομένων. Είναι πάρα πολύ προβληματική η κατάσταση αυτή, αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε σε τόσες λεπτομέρειες με ε, ποσοτικά στοιχεία. Για τα άλλα, συμφωνώ στις υπόλοιπες τροπολογίες, σίγουρα θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Στην τροπολογία 44, 61 και 55 γίνεται λόγος για ειδικά μοντέλα. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να αναφέρουμε συγκεκριμένα μοντέλα, τρόπους διαχείρισης και λειτουργίας, γιατί ε, διεθνώς υπάρχουν και άλλα που δεν αναφέρονται και ίσως στο μέλλον να προκύψουν και νέα. Η επιχειρηματολογία όμως είναι πολύ καλή. Στην τροπολογία 46 η κυρία Ντελή ομιλεί για ένα πενταετές, έτσι πιο μακροπρόθεσμο διάστημα αξιολόγηση. Εγώ είχα προτείνει τριών έως πέντε ετών. Εδώ λέει ένα πλαίσιο πέντε τουλάχιστον ετών. Εγώ προτιμώ τη δική μου διατύπωση. Και άλλες τροπολογίες, η 37, η 38, η 50 και η 51, είναι κάποιες τροπολογίες που συμφωνούμε επί της ουσίας και μπορούμε να καταλήξουμε, πιστεύω τελικά. Όταν μιλάμε για κυρώσεις όμως, πρέπει να ξέρουμε τι εννοούμε. Στην τροπολογία 54, επίσης δεν μου αρέσει η διατύπωση για τις αμοιβέ και τα μισθολογικά κτλ. 56, 57, εντάξει, 58 είναι παρόμοιες με τη δική μου τροπολογία 6. Έχουμε μετά την τροπολογία 59 της κυρίας Ντελή, η οποία ε, ομιλεί για μεταβλητές συνιστώσεις αμοιβών. που να αντιπροσωπεύει το 80% τουλάχιστον των συνολικών αμοιβών τολμώ να αμφισβητήσω τα στοιχεία αυτά, τα αριθμητικά. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να βάλουμε τόσο συγκεκριμένα νούμερα, αλλά είμαι πρόθυμος να το συζητήσω. Η τροπολογία τώρα 60, λέει, η Αρίκ και Τσίμερ λένε ουσιαστικά το ίδιο. Και η 62 αμιλεί επίσης για την πενταετία. Εγώ θέλω να λέω τουλάχιστον τρία έτη, τρία με πέντε έτη, δεν θέλω το πενταετία. Ε, το 63 το ίδιο. Αυτά έτσι επιτροχάδι οι τροπολογίες. Και ελπίζω ε, την άλλη εβδομάδα να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε την επόμενη ή την μεθεπόμενη εβδομάδα για να ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Πριν δώσω το λόγο σε επόμενου ομιλητέ να υπενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής ότι η έκθεση που μας παρουσίασε η Eurofound για την ε, υπηρεσία του Δουβλίνου αναφέρει για δεύτερη φορά την κατάσταση των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε ευρωπαϊκή κλίμακα και κάθε φορά γίνεται ανάλυση ανατομέα. Υπάρχει και μία ανάλυση για το χρηματοπιστωτικό τομέα, φυσικά. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση θα μπορούσε να είναι μία πηγή στοιχείων για να συνεισφέρουμε σε αυτή τη συζήτηση. Παρότι αυτή έρχεται μετά την κατάθεση των τροπολογιών, νομίζω ότι για να βρούμε συμβιβασμούς θα μπορούσαμε να ανατρέξουμε σε πηγές ε, που είναι πάρα πολύ αναλυτικές ε, και που υπάρχουν ε, σε αυτή την έκθεση και που είναι σημαντικές για τη συζήτησή μας. Η κυρία Μέσνερ και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ εξ ονόματο των Φιλελευθέρων και του Γιώργιου Κρόιτσμα να σα ευχαριστήσω που είναι σκιώδη ηγητή και δυστυχώ κολλείται γιατί είχε σημαντικέ ανηλυμένε υποχρεώσει στην εκλογική του περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή για την έκθεσή του. Συμφωνεί η ομάδα μα σε γενικέ γραμμέ μετά όσα είπε και ο κύριο Κρίστενσεν. Γι' αυτό δεν κάναμε δικέ μα τροπολογίε. Και... Ε, συμφωνήσαμε με τις τροπολογίες του κυρίου Τόμας Μαν. Δυσκολίες όμως έχουμε εμείς ως ομάδα και ο κύριος Κρόιτσμαν με τις τροπολογίες ε, των Πρασίνων και της γοέ διότι Νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ περιοριστικές οι προτάσεις τους για τις αμοιβέ των στελεχών και δεν συμφωνούμε καθόλου ως ομάδα. Αυτή τη σύντομη δήλωση προς το παρόν έχω να κάνω, μια που απουσιάζει και ο σκιώδης ηγητή. Βεβαίως όμως είμαστε στη διάθεσή σας και ο ίδιος ε, για τις μελλοντικές συζητήσεις και συνεννοήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξαναπώ στον Όλε Κρίστιας ότι αγαπητέ όλοι οι εκθέσεις σου πάντα είναι πάρα πολύ καλές και συμφωνούμε και εδώ. Τρεις ε, τροπολογίες έκανα και είπες εσύ ότι μπορείς ε, να συμφωνήσει. Στη ότι πολύ καλά είχαμε συνεργαστεί. Θυμήσου, ε, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αυτή. Είναι σημαντικό να λέμε ότι οι τράπεζες καλό είναι καμιά φορά τηρούν και τα όσα υπόσχονται. Είπαν εντάξει, ότι έχουμε ένα κώδικα δεντολογία, δεν είμαστε φιλανθρωπικά ιδρύματα, το κατανοούμε αυτό, αλλά ε, δρούμε και λειτουργούμε μέσα σε μια κοινωνία με ευθύνη. Και πώ θα το πετύχουμε αυτό. Ε, είπε όλα ότι έχουν δυσκολίε οι τράπεζες ε, στη Δανία και αλλού, με πτωχεύσεις, με ανεπαρκή προστασία των αποταμιεύσεων, των καταθέσεων και πώ μπορούμε εμεί να ανατρέψουμε αυτές τις τρευλέ εξέλιξεις, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους καταθέτες να τους προστατεύουμε. Ε, ποια δυνατότητα έχουμε να φέρουν ευθύνη και τα στελέχη των τραπεζών, να ξέρουν τι προϊόντα, τι παράγωγα πουλάνε, τι προσφέρουν στους πελάτες. Και γιατί τα πουλάνε, για να πάρουν ένα καλό πριμ χωρίς να ξέρουν καν τι προϊόντα είναι αυτά, τι παράγωγα. Πολλέ φορές είχαμε διάφορα καλάθια με τοξικά ομόλογα και οι ίδιοι οι υπάλληλοι των τραπεζών που τα πουλούσαν δεν είχαν ιδέα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουν ε, και να ε, έχουν επαφή με την πραγματικότητα και τα στελέχη που έρχονται σε επαφή με καταθέτες και με αποταμιευτές. Για να ανακτήσουν λοιπόν την αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη οι τράπεζες θα πρέπει να λένε σας προσφέρουμε κάποια προϊόντα ε, με στόχο βέβαια το κέρδος αλλά έχουμε και την ευθύνη για αυτά. Ελπίζω και το Συμβούλιο ε, να τα έχει αυτά υπόψη, γιατί, όπως και για τη σταθερότητα τη νομισματική. Αυτή η τροπολογία που λέει ότι ε, τα ηγετικά στελέχη των τραπεζών παίρνουν 300 φορές περισσότερες αμοιβέ από ε, τους υπαλλήλους. Τα ξέρουμε αυτά, δεν χρειάζεται να βάλουμε ε, σε τροπολογία. Είναι λίγο διατύπωση καφενείου, δεν είναι επίπεδου τροπολογίας αυτή. Και σε εποχής, εποχές ε, κρίσεων πάντα συζητούσαμε για τις τράπεζες και στο παρελθόν. Τι, ποιο ρόλο έχουν, ποιο έλεγχο, ποια εποπτεία ε, μπορούμε εμείς να ασκήσουμε ως πολιτικοί. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά και θα πρέπει να τα λέμε και στην Επιτροπή που ασχολείται με την αντιμετώπιση της κρίσης. Γιατί τελικά η κρίση δεν είναι μόνο τραπεζική ή οικονομική, είναι και κρίση των κοινωνικών συστημάτων γενικότερα. Και χαίρομαι που συμμετέχει και η δική μας Επιτροπή σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλε, τελικά πιστεύω ότι θα είναι καλός συμβιβασμό και θα μας ικανοποιεί όλους. Euh, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κυρία Έντμερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί στην ε, ομάδα μεταρρυθμιστών και συντηρητικών θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση είναι παράδειγμα μια πασίγνωστη ε, δοξασία τη Ευρώπη ε, ότι οποιαδήποτε κρίση φτάνει στην πραγματικότητα είναι δικαιολογία για να συγκεντρώνεται στις Βρυξέλλες μεγαλύτερη εξουσία και να αφαιρείται από τα κράτη-μέλη. Είτε είναι φυσική καταστροφή, είτε είναι οικονομική καταστροφή, πάντα είναι μια δικαιολογία, ούτω ώστε να αυξάνουμε την χείρα των Βρυξελών ε, εις βάρος της εξουσίας των εθνικών κυβερνήσεων. Είναι, είναι λάθος, δεν είναι σωστό αυτό. Και πολλέ από τι προτάσει ε, που υπάρχουν και στι τροπολογίε είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν. Να σα δώσω ένα-δύο παραδείγματα. Παραδείγματο χάρη τροπολογία 4. Εκεί ζητάμε ανεξάρτητη επιτροπή για τις αποδοχές. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα 27 κρατημένα να ελέγξουμε αυτές τις ανεξάρτητες επιτροπές. Στην ε, τροπολογία 9 θέλουμε οι υπάλληλοι των ε, τραπεζών να μην κάνουν αντιστάθμιση των κινδύνων σε ιδιωτικό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Και νομίζω ότι είναι και παρίσφρηση στις ιδιωτικέ αποφάσεις του καθενό. Είμαστε αντίθετοι λοιπόν. Θεωρούμε ότι αυτό προτείνεται εδώ είναι όχι μόνο ένα συμπίλημα περί των ε, εξουσιών στις Βρυξέλλες, αλλά είναι και μια μεταφορά αρμοδιοτήτων και ε, εξουσιών, χωρίς μεταφορά όμως και ευθυνών παράλληλα. Και αυτό ε, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Μια διαίρεση, δηλαδή μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες. Λάθος δεν το υποστηρίζουμε λοιπόν. Θέλει κανένα άλλο το λόγο. Η Κομισιόν ίσως. Κύριε Βόλτερ, δεν είναι εδώ. Θα δώσω ξανά το λόγο στον εισηγητή μας τότε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Είμαι πεπισμένος ότι θα καταλήξουμε τελικά σε ένα καλό συμβιβασμό. Χαίρομαι και όλες που διαφωνεί ο κύριος Χέλμερ. Αλλιώς θα άρχιζα να αμφιβάλλω και θα είχα ανησυχίες. Αν έλεγε ότι συμφωνούσε θα ξανακοίταζα την πρότασή μου και θα ψαχνά τι έκανα λάθος. Ε, δεν ε, επεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρυθμίσει τον κλάδο, ξέρετε. Ο κόσμος όλος θέλει να φροντίσει να μην επαναληφθεί αυτή η χρηματοπιστωτική κρίση. Ξέρετε και στι Ηνωμένε Πολιτείε ασχολούνται με το θέμα αυτό και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό τον καιρό προσπαθούν να ρυθμίσουν έτσι την κατάσταση. και για τις αποδοχές και για ε, τις ε, αμοιβέ γενικότερα και ελπίζω και οι η ω να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ευρώπης. Λοιπόν, καλή συνεργασία και προσβλέπω σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Euh, Ευχαριστώ. Έχετε μέχρι τις 16 ε, Μαρτίου προθεσμία. Στις 16 ή 17 θα ψηφίσουμε μάλλον στις 17, για να ετοιμάσουμε την γνωμοδότησή μας πριν η αρμόδια επιτροπή, δηλαδή η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, αποφανθεί που θα γίνει στις 27 Απριλίου. Έτσι. Τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της μεσίας διάταξης και δυστυχώς θα αναγκαστώ να σας προσκαλέσω στο καφέ ή να βγείτε, εν πάση περιπτώσει, λίγο για να κάνετε κανένα τηλεφώνημα, γιατί θα πρέπει μέχρι τις 10.30 να σταματήσουμε τις εργασίες μας. Στις 10.30 θα ψηφίσουμε τις δύο επιστολές για το Ταμείο ε, Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Σταματάει η συνεδρίαση μέχρι τις 10.30.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 so so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

ώστε να μπορέσουμε να συνεχίζουμε αδιακοπτά, αδιάλειπτα. Ε, Όπω ξέρετε, σε λίγο θα ακούσουμε τον Επίτροπο. Είχαμε προβλέψει στι 10.30 την, παρουσία, την ψηφοφορία. Δεν θέλω να αλλάζω την ώρα τη ψηφοφορία, ούτε κι εσεί. Και έχουμε να συζητήσουμε για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Να τονίσω μόνο τον Επίτροπο ότι ίσως κάποια έδρανα μπορεί να φαίνονται αδιανά, αν και υπάρχουν πολύ ικανά μέλη του ΕΛΚΑ που είναι εδώ γιατί αυτό οφείλεται στο ότι το ΕΛΚ κάνει ένα σεμινάριο στη Βουδαπέστη. Ορίστε. Στην πόλη σας. Φαντάζομαι θα το συγχωρήσετε αμέσως. Φτάνουμε λοιπόν να δούμε στην ημερησία μας διάταξη. Έχουμε ένα πρώτο, μια πρώτη επιστολή που την απευθύνουμε στον Αλέν Λαμασούρ που είναι πρόεδρος της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμού και πρόκειται για μια υπόθεση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στο πλαίσιο της ε, βιομηχανίας επίπλωσης και υφαντουργίας και ένδυσης της Λιθουανίας. Μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ. Και contre. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ομόφωνα. Ομαδοποιήσαμε την ψήφο γιατί ήταν δύο υποθέσεις της Λιθουανίας. Τέλος λοιπόν με τις ψηφοφορίες. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την υπομονή του και με τα χαράς να τον καλωσορίσω επισήμως ε, στη, υπό την ιδιότητά του ως Επιτρόπου. Ξέρετε, έχουμε μια κακή συνήθεια εδώ πέρα. Θέλουμε να σας βλέπουμε συχνά. Για να είμαστε βέβαιοι πως ε, είμαστε συγχρονισμένοι με τις αναλύσεις και με τα θέματα που εξετάζουμε. εξετάζουμε την υπόθεση της στρατηγικής 2020. Ε, είναι πολύ σημαντικό για μας να σας ακούσουμε την επάβρη της παρουσίασής σας και σας δίνω αμέσως το λόγο για να μας πείτε ποια είναι, είναι, ποιοι είναι οι βασικοί προσανατολισμοί και έπειτα ε, θα έχετε τη χαρά να υποστείτε μια σειρά έρωτα απαντήσεων. Φαντάζομαι πως ήδη θα έχετε συνηθίσει σε αυτή τη διαδικασία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας συναντήσω. Η πρώτη συνάντηση από την ανάληψη των καθηκόντων της Νέας Επιτροπής και είναι η πρώτη ευκαιρία που είχα να σας συναντήσω ε, γιατί την τελευταία φορά συναντήθηκαμε υπό άλλες συνθήκες και ξεκινάμε με ένα κρίσιμο έγγραφο. Είμαι έτοιμος να το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά όπως είπε και η Πρόεδρος, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω και κάθε ευκαιρία που έχουμε για να συζητήσω με τους ε, βουλευτές ε, της Επιτροπής σας και ακόμα και διμερός ε, και διαπροσωπικά αλλά και στην Ολομέλεια για να συνεχίσουμε το διάλογο. Γιατί το θέμα είναι κρίσιμο, ιδίως μέσα σε συνθήκες κρίσης. Χθε η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για έξυπνη, πράσινη και συνολική ανάπτυξη. Και νομίζω ότι μια στενή συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν είναι σημαντική για την επιτυχία αυτής της στρατηγικής. Ε, δέκα χρόνια μετά από τη στρατηγική της Λισαβόνας έρχεται αυτό το κείμενο και τελειώνει φέτο αυτή η περίοδο της δεκαετία. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πω η στρατηγική για να καταστήσουμε τη στρατηγική τη Λισαβόνα θα πρέπει να είναι πιο απλή, πιο αποτελεσματική αλλά και πιο εστιασμένη. Κατά την άποψή μου αυτό το έγγραφο υλοποιεί αυτού του στόχου και υλοποιεί δύο σημαντικού ε, στόχου. Ο ένα είναι βραχυπρόθεσμος, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε δηλαδή την ε, τρέχουσα οικονομική κρίση και να δώσουμε ξανά δουλειά στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτό. Μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να κατευθύνει το οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο της Ένωσης προς μια κατεύθυνση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις, οι τεχνολογικές, δημογραφικές και κλιματικές των, της αλλαγής. Η, Λισαβόνα, η ατζέντα της Λισαβόνας Ήδη είχε προναγγείλει αυτό και η νέα στρατηγική θα πρέπει να δώσει αποτελέσματα στην, στα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Η πρότασή μας θέτει την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας στο κέντρο της προσπάθειάς μας, ακριβώς όπως το θέλουν και οι ενδιαφερόμενοι. Ε, νομίζω ότι είναι η το βασικό μέλημα όλων των Ευρωπαίων σήμερα. Οι στατιστικές είναι πολύ σοβαρές, ε, γιατί η ανεργία στην Ευρώπη είναι περίπου στο 10% του εργατικού δυναμικού και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω. Μετά από την μείωση της ανεργίας, που είναι το πιο βασικό θέμα, είναι το μεσοπρόθεσμο ο μεσοπρόθεσμος συγγνώμη, στόχος, ε, καλύτερες θέσεις απασχόλησης και κοινωνική ένταξη. Η Κομισιόν έχει, προβλε... έχει προβλέψει τρεις προτεραιότητες, ε, οι δηλαδή φορείς της ανάπτυξης, που είναι και οι πυλώνες αυτής της στρατηγικής. Και είναι Πρώτον, ε, έξυπνη ανάπτυξη, να αναπτύξουμε μια οικονομία που να βασίζεται στην γνώση και στην καινοτομία. Δύο. Βιώσιμη ανάπτυξη, προωθώντα ε, μια πιο πράσινη, πιο αποτελεσματική, με καλύτερη χρήση των πόρων και πιο ανταγωνιστική ε, οικονομία. Τρίτον, ανάπτυξη συνολική, με μια οικονομία πλήρους απασχόλησης, με κοινωνική και οικονομική και εδαφική συνοχή. Αυτά είναι σημαντικά. Η πλήρης ανάπτυξη. Βασιζόμαστε στην στρατηγική απασχόληση και στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία. Θα συμφωνήσετε ότι πρέπει να εντάξουμε τις κοινωνικές πολιτικές και το κάνουμε αυτό με αυτή τη στρατηγική πιο πολύ από ότι με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Και αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τους στόχους που μας ενδιαφέρουν και οι πολιτικές ε, σε άλλους τομείς θα πρέπει τους κοινωνικούς στόχους και την απασχόληση να τους ε, λαμβάνουν επίσης υπόψη. Επίσης, υπάρχει μια βασική κοινωνική ε, συνιστόσα στον πυλώνα για την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν περιορίζεται δηλαδή μόνο στον τρίτο πυλώνα. Η βελτίωση της εκπαίδευσης, της διαβίου κατάρτισης Αυτά είναι σημαντικά για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόληση. Να βελτιωθούν οι σχέσει μεταξύ τη θέση, απασχόληση, η σχέση μάλλον μεταξύ των θέσεων απασχόληση και τη εκπαίδευση για να δημιουργηθούν γέφυρε για του νέου. Και αν έχουμε και μια ανταγωνιστική οικονομία, αυτό θα έχει θετική επίπτωση στην αγορά εργασία μέσω τη δημιουργία φερρυπίν πράσινων θέσεων απασχόληση. Αυτό αρχίσαμε να συζητούμε και με τον Επίτροπο για την Κλιματική Αλλαγή. Με την Επίτροπο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, ε, το κέντρο της στρατηγικής αυτή θα είναι οι στόχοι. Θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος για να υλοποιηθούν οι τρεις ε, ε, προτεραιότητες. Έχουμε τρεις πυλώνες και πέντε στόχοι. Θέλουμε λιγότερους σαφείς κατανοητούς στόχους που θα βασίζονται σε κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής και αυτά να τα καταστήσουμε πιο ορατά μέσω της συζητήσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, η Κομισιόν δίνει σημασία στις κοινωνικές πολιτικές και στην πολιτική απασχόλησης. Και αυτό ε, δείχνει με το στόχο της απασχόλησης ότι αυξάνεται η απασχολησιμότητα του πληθυσμού, ε, μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών από το 69% σε τουλάχιστον 75%. Δεύτερο σημαντικό κοινωνικό στόχο είναι ε, η μείωση του ποσοστού των Ευρωπαίων ε, ε, κατά 25% που ζουν κάτω από το όριο φτώχεια, δηλαδή να φύγουν, να βγάλουμε από τη φτώχεια 20 εκατομμύρια ανθρώπου. Τρίτον, εκπαίδευση, να μειωθούν ως από το 15% στο 10% οι άνθρωποι που φεύγουν νωρίτερα από το σχολείο. Και Ξέρουμε ότι αυτοί οι στόχοι μπορούν να υλοποιηθούν μέσω στρατηγικών που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Η ποικιλομορφία είναι ευρωπαϊκή αξία. Θα πρέπει όμως την ποικιλομορφία να τη θεωρήσουμε και ως πρόκληση. Ορισμένοι πρέπει να σκαρφαλώσουν πιο απότομους ε, πιο απότομες κλήσεις, πιο, ε, πιο δύσκολα βουνά. Γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, από πού ξεκινάει το κάθε κράτος μέλος. Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη για να καθορίσουν τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι ελπίζουμε να είναι και ρεαλιστικοί αλλά και φιλόδοξοι. Πιστεύω ότι και οι στόχοι της Κομισιόν είναι φιλόδοξοι και ρεαλιστική. Προτείνουμε μια θεματική προσέγγιση, ώστε τους πέντε στόχους να τους προωθήσουμε μέχρι πρωτοβουλίες. Έχουμε τρεις πυλώνες, πέντε στόχους. Ε, τρεις από αυτούς είναι, σχετίζονται με τις κοινωνικές πολιτικές και, τους, και την απασχόληση. Καταρχάς η ατζέντα για τις νέες δεξιότητες και, τις, και την την εργασία. Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της ε, εργασίας. Υπό την ατζέντα ε, αυτή η βασική στρατηγική είναι η flexicurity, η ευέλικτη ασφάλεια. Είναι σημαντική για να εκμοντερνιστεί η αγορά εργασίας, να υπάρξει συνένεση που έχει ε, προκύψει τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει ευελιξία αλλά και ασφάλεια της απασχόλησης. Η flexicurity θα πρέπει να μας βοηθάει να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες που τη χρειαζόμαστε, να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα στην εργασία μας και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Γι' αυτό η Κομισιόν θα αναπτύξει περισσότερο τα νέα, τα νέα προγράμματα. Ε, αυτό σημαίνει ότι θα δούμε τι δεξιότητες χρειάζονται σε κάθε θέση απασχόλησης. θα βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους να μπουν στην αγορά εργασίας θα συμφιλιώσει την ε, εργασιακή ζωή και την ε, οικογενειακή ζωή και θα προωθήσουμε μια μεγαλύτερη επαγγελματική καριέρα, μακρύτερη επαγγελματική καριέρα. Ε, η δεύτερη επικοινωνία της Κομισιόν για τις νέες δεξιότητες για νέες δουλειές θα δώσει απαντήσει σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, ανάπτυξη μιας πλήρους ατζέντα για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης και οι επιδόσεις των νέων στην αγορά εργασία. Εδώ θα παρουσιάσω ένα πλαίσιο δράσης ολοκληρωμένο για να διευκολύνουμε την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Θα βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ της εκπαίδευσης και της δουλειάς. Αυτό είναι πολύ βασικό σε αυτό το επίπεδο. Οι νέοι θα αντιμετωπίσουν όλο και το περισσότερο ε, δυσκολίες μετάβασης στην αγορά εργασίας. Χρειάζεται δράση λοιπόν για να προωθήσουμε την μαθητεία, τα στάζ, ε, την επαγγελματική εμπειρία ε, παράλληλα με, την, με τις συμβουλές προς τους νέους. Θα θυμάστε ότι όταν σας συνάντησα στην ακρόασή μου τον Ιανουάριο εδώ στο Κοινοβούλιο ε, ήμουν υπέρ της ιδέας ε, ενός ε, σχήματος ανάλογου με το Erasmus για την πρώτη δουλειά για τους νέους, ούτως ώστε να αποκτήσουν έτσι, ευκαιρίες οι νέοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. και πιστεύω ότι αυτό το νέο πρόγραμμα θα δρομολογηθεί πολύ γρήγορα. Θα υποστηρίζει τοποθέτηση των νέων ε, ενός κράτους μέλος ε, που θα βρίσκουν θέση σε μία, σε μία άλλη χώρα. Το τρίτο σημείο είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα εναντίον της ε, φτώχειας που θα αυξήσει σημαντικά την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης με ορίζοντα το 2020. Μαζί με το στόχο της μείωσης της φτώχειας θα εντείνει την ε, έμφαση της στρατηγικής στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, στην κοινωνική ένταξη και στην κοινωνική προστασία και ιδίω ε, θα δοθεί ένας μεγαλύτερος ρόλος στην παρακολούθηση της πρόοδου. Κυρία Πρόεδρε, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ε, στρατηγική για το 2020 θα είναι πολύ σημαντικό. Η Κομισιόν θέλει το Κοινοβούλιο να δώσει τη γνώμη για τις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τι ολοκληρωμένε κατευθυντές γραμμές. Τα Εθνικά Κοινοβούλια επίσης θα πρέπει να εμπλακούν περισσότερο και να συμμετάσχουν σε αυτή τη στρατηγική του Ευρώπη 2020. Επίσης, οι περιφέρειες και οι τοπικέ αρχές ε, θα πρέπει να εμπλακούν και να υπάρχει μεγαλύτερη σχέση με τις προτεραιότητε που θέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τις εθνικές στρατηγικές, ε, τους, ε, τις δαπάνες και τα προγράμματα. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να εμπλακεί πιο πολύ στο σχεδιασμό των πολιτικών καθώς και της εφαρμογής τους. Μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που θα πρέπει να συνδεθεί με, την, ε, με τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 θα μπορούσα να συνομιλήσω με τα μέλη της Επιτροπής για να συζητήσουμε τις πολιτικές που είναι υπό την ευθύνη μου. Μεταξύ των βασικών πολιτικών για το εγγύς μέλλον είναι η εξή. Δεξιότητες και απόκτηση ε, δεξιοτήτων για τις μελλοντικέ ανάγκες. Flexicurity, ευελίξη ασφάλεια. Ε, συμμετείχα σε αυτό το σεμινάριο που οργανώθηκε τον κύριο Σάρκας χθες ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνάντηση αυτή, ε, ο διάλογος, μου έδωσε πολλές ιδέες, ε, μας ενέπνευσε. Η πραγματική ενεργή ένταξη, πράσινες θέσεις απασχόλησης και πρασίνισμα της οικονομίας. Ξέρω ότι η Κομισιόν σας, η Επιτροπή σας δουλεύει για πολλές από αυτές τις εκθέσεις και περιμένουμε με υπομονεσία να ακούσω τις απόψεις σας. Το θέμα είναι λοιπόν η στρατηγική Ευρώπη 2020. Πού μας πηγαίνει έτσι όπως εκδόθηκε, έτσι όπως παρουσιάστηκε από την Κομισιόν. Θα ξέρετε ότι το ερεινό Συμβούλιο στις 25 και 26 Μαρτίου θα συζητήσει την πρόταση της Κομισιόν. Βάσει αυτών των συμπερασμάτων, η Κομισιόν θα παρουσιάσει ε, μια πιο λεπτομερή πρόταση για τις ε, σωματωμένες κατευθυντήριες γραμμές, ε, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για την απασχόληση που βασίζονται στη συνθήκη. Θα ξανασυναντηθούν αυτά στο Συμβούλιο ε, με βάση τη γνωμοδότηση του ε, Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο του Ιουνίου θα επικυρώσει αυτή τη στρατηγική. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, πιστεύω στεναρά ότι η επιτυχία της νέας στρατηγικής είναι ζωτική σημασία για τη μελλοντική ευημερία και το πλούτο των λαών της Ευρώπης. Αν θέλουμε ε, η πυρός μας να εξακολουθήσει να είναι ηγετική ε, οικονομία και κοινωνικό μοντέλο ε, που θα προωθεί την ευημερία των λαών της, θα πρέπει όλοι να συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια για να επιτύχει. Ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός σε αυτή τη διαδικασία. Περιμένω πραγματικά με ανυπομονησία να συζητήσουμε, να συνεργαστούμε για να καταστήσουμε αυτή την ε, στρατηγική μια πραγματική επιτυχία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Τώρα έχω το δίλημα της Προέδρου. 17 συνάδελφοι ζητούν το λόγο και θα εφαρμόσω το φοβερό κανόνα της Προέδρου. Δύο λεπτά έκαστος για να μπορέσουν όλοι να μιλήσουν και μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο όχι στο τέλος για να μην απαντήσει μόνο στις ερωτήσεις που θέλει και σε καμία άλλη αλλά θα ακούμε τρεις παρεμβάσεις και μετά θα δίνουμε το λόγο Κλείνει όμως ο κατάλογος των ομιλητών έτσι Α, συν τρεις, είκοσι σύνολο, ωραία Ρίσαρτ Φάρπ και μετά οι υπόλοιποι. It was my phone. Α, το κινητό μου ήταν. Birds. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Η στρατηγική της Λισαβόνας κατέληξε ε, φιάσκο σκέτο. Δεν ε, κατάφερε να καλύψει κανένα στόχο της. Ένα σλόγγαν ήταν ε, περισσότερα και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Και καταλήξαμε να έχουμε και λιγότερες και χειρότερες. Η στρατηγική για το 2020 είναι καλύτερη από τη στρατηγική της Λισαβόνας γιατί είναι και πιο σύντομη και έχει και λιγότερους στόχους. Αλλά από άλλε πλευρές ευκολόγιο είναι και αυτή, όπως ήταν και η στρατηγική τη Λισαβόνα. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν με θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τι είδου θέσει απασχόλησης. επισφαλή. και πού είναι η ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, ποιο συντονισμό. Τα κράτη-μέλη κάνουν ό,τι θέλουν δεν έχουν ε, επιθεωρήσεις εργασίας σωστές με την απαραίτητη στελέχωση και το προσωπικό που χρειάζονται για να κάνουν ελέγχους. Στη χώρα μου επικρατεί δουλεία. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες. Οι λεγόμενοι αυτοαπασχολούμενοι ή οι πραγματικοί αυτοαπασχολούμενοι έχουν και αυτοί προβλήματα. Συνδικάτα, ποια συνδικάτα, τι συνδικαλιστικές οργανώσεις μπορείτε να έχετε ε, όταν είναι τόσο επισφαλείς οι ε, μορφές εργασίας και οι θέσεις απασχόλησης. Εκπαίδευση, κατάρτιση, ποια κατάρτιση. Οι περισσότερες θέσεις αυτές είναι ανειδίκευτες, χειρονακτική εργασία. Δύο μέρες εκπαίδευση χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πολύ εργαζόμενοι στη χώρα μου ε, και πολλοί κόσμοι γενικά ε, δεν δηλώνει ότι είναι ε, από αυτούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γιατί το θεωρεί εμπόδιο ότι δεν θα βρει δουλειά. Flexicurity, ευελιξ ασφάλεια, υπάρχει μόνο στη Δανία. Αυτοί έχουν συνδυάσει την ευελιξία με την ασφάλεια. Αλλά πουθενά άλλου δεν λειτουργεί αυτό το σύστημα. Είναι χήμερα, απάτη, ψέμα. Και το 2020 είναι απλώς ένα όνομα, μια ιδέα, δεν είναι τίποτα ουσιαστικό. Η κυρία Λίν, ευχαριστώ και σας καλωσορίζω κύριε Επίτροπη. Ε, σε κάποιο βαθμό συμφωνώ και εγώ ότι δεν επέτυχε όλους τους στόχους της η, συγγνώμη, διαδικασία της ε, Λισαβόνας. Και τώρα έχουμε φτάσει στο κείμενο 2020. Μιλήσατε για την καταπολέμηση της φτώχειας και στο έγγραφο το λέτε. Χαίρομαι που γίνεται λόγος για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, από ότι το αρχικό έγγραφό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί φοβήθηκα ότι θα μας είχε απορροφήσει η χρηματοοικονομική κρίση και ε, δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με τα υπόλοιπα. Είπατε ότι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η κοινωνική ένταξη συγγνώμη, ε, συνδέεται με την καταπολέμηση στόχιας. Αλλά Πού εντάσσεται η στρατηγική του 2020. Ξέρω ότι η πρόεδρος γελάει γιατί πάντα μιλάω για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Ναι, θα συνεχίσω να το κάνω. Επίσης, ε, για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Ε, φοβάμαι ε, ότι θα μείνει εκτός εξίσωσης και θα το, θα το παραπετάξει και η Κομισιόν και το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο. Με ανησυχεί λοιπόν αυτό. Και το άλλο θέμα, οι στόχοι. Με βάση αυτό που συνέβη, που δεν συνέβη στη Λισαβόνα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι στόχοι θα υλοποιηθούν. Γιατί πολύ ωραία να έχουμε ωραία συναισθήματα, να λέμε ότι θέλουμε να τα, να υλοποιήσουμε όλα αυτά, να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ε, να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη, αλλά πώς θα επιτευχθεί αυτό. Και για να πάω τώρα στην ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Στο έγγραφο λέτε ότι θα μετασχηματίσετε την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού. Θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο πώς θα λάβει χώρα αυτός ο μετασχηματισμός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε ακόμα δύο ανθρώπους. Πρώτα τον κύριο Σάρκας και μετά τον κύριο Μάνα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε. Ε, σας ευχαριστώ που παραστήκατε χθε ε, στο σεμινάριό μας. Ε, βλέπω ότι κάνετε μια προσπάθεια να πλησιάσετε το Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ για τα αρχικά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αλλά κρίμα που τα λόγια σας δεν εντάσσονται και στο κείμενο. Ε, Καλύτερες απασχόλησης πουθενά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει πολιτική κοινωνική ένταξη. Φοβάμαι, κύριε πίτροπε, ότι αυτό το έγγραφο, ε, τουλάχιστον για μας τους σοσιαλιστές, βρίσκεται κάτω από τις προσδοκίες μας. Αυτό που είναι πολύ πιο σοβαρό, είναι πολύ πιο κάτω από τις προσδοκίε των Ευρωπαίων. Ε, ίσως δεν έχει γίνει επαρκής ανάλυση. Ίσως θεωρείτε ότι Αντιμετωπίσει μια κρίση σε επίπεδο ανάπτυξης. Όχι, είναι ε, κρίση για την απασχόληση, κρίση οικολογική, κρίση σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι θεωρείται ότι αν θα βελτιωθεί η οικονομία, αυτόματα θα βελτιωθούν και όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Θα εξαλειφθούν. Όχι. Δεν λύνονται αυτόματα τα προβλήματα κοινωνική ένταξη, τα προβλήματα έλλειψη κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει καμία πολιτική φιλοδοξία στο κείμενό σα. Τίποτα δεν ακούσαμε. Ακούτε μόνο του ε, γραφειοκράτε και τους υπάλληλου. Δεν ακούτε αυτά που λένε οι πολίτες, δεν ακούτε αυτά που λένε τα συνδικάτα, δεν ακούτε αυτά που λένε οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε απάντηση στο, στην ουσία του προβλήματος, στην απαρχή του προβλήματος. Ε, μιλάμε για την χρηματοπιστωτική κρίση, μια τρελή κρίση που, κα, που κατέστρεψε την οικονομία, κατέστρεψε χιλιάδες ε, θέσεις απασχόλησης. Ε, αλλά, πρόεδρε, ε, αλλά Επίτροπε, η απάντηση δεν είναι η οικονομική ανάπτυξη που θα λύσει όλα τα προβλήματα. Θέλουμε μια πραγματική στρατηγική που θα τα εξορροπεί όλα. Τα πολιτικά, τα οικολογικά, τα κοινωνικά, τα οικονομικά. Ε, και με τι εργαλεία. Δεν έχουμε εργαλεία. Ελπίζουμε να μα δοθούν απαντήσει επόμενου μήνε. Τόμας Φαν, ευχαριστώ. Ε, και ευχαριστώ και τον Επίτροπο που ήρθε τόσο νωρί. Δεν μπορώ παρά να απαντήσω στον κύριο Σέρκα ότι υπήρξε ένα έγγραφο εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής 24 Νοεμβρίου 2009. Συμμετείχαν όλοι και οι κοινωνικοί εταίροι και οι πάντες και μέχρι τι 15 πρώτου έπρεπε να δώσουν τις θέσεις τους. Δεν τελείωσε κενό αέρος λοιπόν, ούτε ουρανοκατέβατο αυτό το έγγραφο. Έχω δύο ερωτήσεις. Ερώτηση πρώτη. Στη Λισαβόνα είχαμε αυτέ τι απώλειε, κύριε Επιτροπή, διότι τα κράτη-μέλη δεν ακολούθησαν δεν ήταν γνωστό στα κράτη-μέλη ποια είναι η ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της ε, ε, προσπάθειας και δεν μπορούσαμε να ε, ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη. Το 2004 ήδη έλεγε η έκθεση ΚΟΚ naming and shaming. Ε, θα κατονομάζονται τα κράτη-μέλη που δεν ε, ανταποκρίνονται και θα ε, διαπομπεύονται. Εγώ είμαι διάπειρο υποστηρικτή αρχή αρχής και ξέρω τι γίνεται στα κράτη-μέλη, ξέρω και τι δεν γίνεται στα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε έτσι περισσότερο να βγούμε προ τα έξω και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Και ένα δεύτερο, σωστά είπατε ότι θα πρέπει να έχουμε στόχους και να ε, ακολουθούν και τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ερωτώ, ποιε είναι οι πιθανότητε που βλέπετε να επιβιώσει το μέλλον και να δημιουργηθεί αυτή η δυνατότητα ε, επιβίωση. Είπαμε, ο στόχο είναι να εγκαταλείπουν όσο γίνεται λιγότερο το σχολείο νωρί. 10% ε, και κάτω του 10% είναι εφικτότατο αυτό ο στόχο. Και χρειάζονται μέτρα όμω. Τα κράτη-μέλη τι κάνουν γι' αυτό. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει εκεί μεγάλη ε, αποστολή. Ε, Μήπω εκεί θα έγκυται και η βιωσιμότητά του στο μέλλον. Thank you Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι με τον κύριο Φέρμπερ διαφέρουμε στην αξιολόγηση της στρατηγικής της Λισαβόνας. Δεν ήταν απόλυτα επιτυχής βέβαια, αλλά νομίζω πως είναι άδικο να λέει κανείς πως ήταν απόλυτη αποτυχία. Επειδή προέρχομαι από μια συγκεκριμένη περιφέρεια, γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι τα μειονεκτήματα της μακροπρόθεσμης, ε, του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και πώς και γιατί απέτυχε σε πολλές ε, περιπτώσεις ένα διαφορετικό βέβαια οικονομικό σύστημα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς ε, προγραμματισμό και σε αυτήν την σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά κάτι τέτοιο θα πρέπει να γίνει γιατί χρειάζεται να θεωρηθεί καταρχήν. Δεύτερον, διότι είναι προφανές ε, πως ορισμένα από τα προβλήματα, ορισμένα από τα διαστατικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας μπορούν μόνο μακροπρόθεσμα να αντιμετωπιστούν. Δεν μπορούν δηλαδή να λυθούν σε ένα ή δύο χρόνια. Χρειαζόμαστε μακρύτερη ε, πιο μακρόπνο μάλλον ε, όραμα για τις μεταρρυθμίσεις και Όντως ε, δεν έχουν επιτευχθεί όλοι οι στόχοι της Λισαβόνας, αλλά ε, δεν είναι δίκαιο να πούμε ότι δεν επιτεύχθησαν καθόλου. Ε, δηλαδή υπήρξε μια αύξηση των ποσοστών απασχόλησης για τις γυναίκες, υπήρξε επίσης ένα, μια δρομολόγηση στον δρόμο προς την ανταγωνιστικότητα. Μετά συνέβη η κρίση. Και είναι προφανές πως η κρίση κατέστρεψε έναν πολύ μεγάλο αριθμό θέσεων που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο και αυτό είναι νομίζω ε, σαφές και ότι δεν αρκεί δηλαδή οι προσωρινέ θέσεις απασχόληση να δημιουργούνται μόνο γιατί αυτέ δεν προσφέρουν ασφάλεια στους εργαζόμενους. Πρέπει λοιπόν να αποκομίσουμε κάποια διδάγματα αλλά να μην τα πετάξουμε όλα μαζί και την αδυναμία της διακυβέρνησης και εκεί νομίζω πως ε, το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 έχει βελτιωθεί εστιάζοντας σε λιγότερους αλλά πιο σημαντικούς στόχους και ενισχύοντας την ε, ιδιοκτησία των κρατών μελών και την δομή διακυβέρνησης για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Βεβαίως το έγγραφο αυτό δεν δημιουργήθηκε στις τρεις εβδομάδες της νέας αυτής επιτροπής. Είχε γίνει προπαρασκευαστική εργασία αλλά η νέα Επιτροπή είχε μια φοβερή δυνατότητα να συζητήσει και να ολοκληρώσει το κείμενο και μπορώ να σας πω ότι είναι από τα κεντρικά σημεία που ε, συζητήθηκαν ήταν η εφικτή και αξιόπιστη στόχη. Τα όσα περιγράψαμε λοιπόν πιστεύουμε πως μπορούν να υποστηριχτούν από τα θεσμικά όργανα και τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, είμαι ευτυχής που η κυρία Λέιν εκτιμά και καλεί την προσοχή στο στόχους ε, και στο κοινό στόχο. Είναι ένα σημαντικό σημείο, είναι ένα νέο στοιχείο. Είναι ένα σχετικά σύντομο κείμενο, οπότε ε, δεν μπορούν να συζητηθούν όλες οι πτυχές αλλά δεν είναι απλό να μιλάμε για μέσους όρους ευρωπαϊκούς. Πρέπει να δούμε και πέρα από αυτούς και όταν δούμε τις ευάλωτες αυτές ε, ε, ομάδες που υπόκεινται σε διακρίσεις θα πρέπει να έχουμε πιο στοχοθετημένα προγράμματα. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το τομέα αρμοδιοτήτων της κυρίας Ρέντινγκ τώρα, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διότι στόχος να χρησιμοποιείται πιο στοχευμένα ακριβώ και πιο αποτελεσματικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να αντιμετωπίσουμε το θέμα του κοινωνικού αποκλεισμού και τη μείωση της ανεργίας που μας απασχολεί και μας ενδιαφέρει. Α, υπάρχει βεβαίως ανάγκη να ενισχυθεί η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού, αλλά και αυτό είναι ένα σχετικά καινούριο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να γίνει μια ε, καλύτερη προσπάθεια συντονισμού όπως είπε και ο κύριος Μαν, αυτός ο συντονισμός θα πρέπει να γίνει υλοποίηση τελικά, όχι να μείνουμε μόνο στο συντονισμό των προσπαθειών. Ευχαριστώ. Επόμενοι ομιλητές. Ο κύριος Τράγιαν Ουρντεοάνου, συγγνώμη, και μετά η κυρία Πλάμ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που μοιράζεστε μαζί μας τις σκέψεις σας. Άκουσα τα πρόσφατα σχόλιά σας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ βασικό και ουσιώδες. Δηλαδή, πώς βλέπετε να συνδυάζεται η ζήτηση και η προσφορά της ε, απασχόλησης και της εργασίας. Με άλλα λόγια, πώς μπορεί κανείς να εγκαταλείπει το σχολείο Και, μάλλον πώς μπορεί κανείς να αποτρέψει τα σχολεία και τις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης να παράγουν μαζικά ανέργους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε ε, για την εισαγωγή σας και για τις ε, δηλώσεις σας. Εγώ έχω να σας κάνω μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Γίνεται λόγος για πράσινη οικονομία, έτσι, και για υφόρο ανάπτυξη και βιώσιμη. Ωραία. Ε, και πράσινες θέσεις απασχόλησης. Σας ερωτώ λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πιστεύετε ότι χρειάζεται ε, ειδική καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής, μια πράσινη λύση. Γιατί το λέω, να σας πω τι εννοώ. Για τη διαβίου εκπαίδευση, lifelong learning, ε, γίνεται λόγος για 8 βασικές δεξιότητες. Θα βάλετε και ένα, τι εδώ τώρα για τη πράσινη ανάπτυξη, για το περιβάλλον. Και ένας από τους στόχους σας που μας προτείνατε είναι μια αγορά εργασίας που να συμπεριλαμβάνει περισσότερες γυναίκες στην αγορά. Και τι θέλει να κάνει γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, νομοθετικό πρόγραμμα για να καταπολεμήσει την ανισότητα και στις αμοιβέ ε, ανδρών και γυναικών. Για να συμμετέχουν πιο πολύ στην αγορά οι γυναίκες. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρή Μαντελή και μετά ο κύριος Ε, κύριε Πρόεδρε, Καλημέρα σας. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, εξαγγείλατε στόχου που μα φαίνονται πάρα πολύ φιλόδοξοι και είπατε μείωση της φτώχεια κατά 20 εκατομμύρια. Η στρατηγική της ε, Λισαβόνας εστέφθη με πλήρη αποτυχία. Εκεί λέγαμε μάλιστα να εκριζωθεί η φτώχεια. Τώρα τα έχουμε μαζέψει λίγο. Αλλά ε, από πού τα βρήκατε αυτά τα στοιχεία, πώς τα αξιολογείτε, πώς τα ποσοτικοποιείτε. Εμείς ε, προτείνουμε να μειωθεί κατά το μισό τουλάχιστον η φτώχεια. Είναι επίγουσα η κατάσταση. Αυτά λένε οι πράσινοι. Μετά, ε, μιλάτε για τους νέους και την ανεργία των νέων. Είπατε ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερη κατάρτιση, εκπαίδευση, μαθητείες, στάζ. Δεν είναι καλή λύση αυτό. Γιατί το στάζι σήμερα οδηγεί στην επισφαλή μορφή εργασίας. Ένας νέος πριν ε, βρει κανονική δουλειά έχει περάσει από διάφορες περιόδους μαθητείας. Και αν δείτε πόσο πληρώνονται οι σταζιέρ είναι ψίχουλα. Ενώ κάνουν κανονική δουλειά, καλύπτουν πάγιες ανάγκες ε, ε, και κάνουν δουλειά υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης δεν μιλάτε για την αυτονομία των νέων. Θα επανέλθετε σε αυτό επίσης και στην ιδέα του κατώτατου ε, εισοδήματο για όλου, ανεξάρτητα από την ηλικία του. Επίση, μιλάτε για τον έρασμο, το Εράσμο. Το Εράσμος δεν είναι προσβάσιμο σε όλου. Οι νέοι ασκούμενοι 16 ετών, α πούμε, θέλουν να πάνε σε μια άλλη χώρα να καλύψουν τον κόσμο, να δουν τι γίνεται αλλού, δεν μπορούν να το πράξουν. Και επίση ο έρασμό δεν είναι μόνο για νέο. όταν κάποιο ε, μεγαλύτερης ηλικίας χάνει τη δουλειά του, γιατί να μην μπορεί ε, να συμμετέχει στο Εράσμος, αν πρόκειται για διαβίου κατάρτιση. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής του δεύτερου γύρου αυτού, ο κύριος Ζόρς Πακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε ε, στο Κοινοβούλιο και λαμβάνετε υπόψη και αυτά που σας λέμε. Θα ήθελα να σας αναφέρω τρία σημεία. Πρώτον, για τις λεγόμενες πράσινες θέσεις απασχόλησης, green jobs. Θέλω να σας ρωτήσω. Έχετε δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, ακριβώς αυτή τη μεταβατική περίοδο ε, από τη μετάβαση, τη μετάβαση από την κλασική βιομηχανία στην πράσινη οικονομία. Πώς θα γίνει αυτό, γιατί χάνει πολύ κόσμο στη δουλειά του. Και δεύτερον, είπατε καλύτερες θέσεις απασχόλησης για να δημιουργηθεί ευημερία για τους πολίτες. Στη στρατηγική 2020 διάβασα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλίνει από τον κανόνα που λέει ότι ε, η εργασία θα είναι μόνιμη και ε, αορίστου χρόνου ή ορισμένου χρόνου εργασία γίνεται ο κανόνας. Το άλλο είναι μάλλον η εξαίρεση. και ε, ο κόσμος αναγκάζεται να ζει από επιδόματα, ανεργίας, επανένταξης μέχρι κάποια στιγμή να βρει ε, κανονική δουλειά και να μπει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και ένα τρίτο για την παιδεία. Είπατε ότι σας απασχολεί ε, ιδιαίτερα η κοινωνία της γλώσσης, η εκπαίδευση, η παιδεία και η πρόθεσή της. Τα ίδια λέει και η Λισαβόνα Δυσκολίε έχουμε τη στιγμή που πρέπει να υλοποιηθούν όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Γενικότερα εκπαιδευτική πολιτική ε, παραμένει ε, πολύ ακόμα στη σφαίρα των κρατών μελών κατά την άποψή μου. Κύριε Πίτροπε. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Πολλές από αυτές τις ερωτήσεις που ακούσαμε σε αυτό το γύρο αφορούν θέματα που είναι συναρμοδιότητα με άλλους επιτρόπους. ξεκινάω από το πρώτο που είναι και το πιο κρίσιμο, το μακροοικονομικό περιβάλλον το μακρονομικό πλαίσιο. Είναι αλήθεια ότι αυτό που εγώ από τη θέση μου μπορώ να υποστηρίξω είναι η πλευρά της προσφοράς της αγοράς εργασίας μέσω καλύτερης κατάρτισης, μέσω ανταγωνιστικής εργατικής δύναμης, μέσω της διαβίου κατάρτισης. Αυτά είναι από την πλευρά της προσφοράς. Αλλά για τη ζήτηση θα πρέπει να συνεργαστώ με τον Όλυ Ρεν, θα πρέπει να δω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τα μακροοικονομικά προγράμματα για τις ε, διάφορες χώρες σε μια εποχή όπου ένας υψηλός αριθμός ε, χωρών έχουν υψηλότατα ελλείμματα. Και τα επόμενα χρόνια θα επιφέρουν ε, μεγαλύτερα, μεγαλύτερη δημοσιονομική λιτότητα. Νομίζω ότι σε αυτό το μακροοικονομικό διάλογο θα πρέπει να θέσουμε και τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα απασχόλησης. Έχουμε κάνει τα πρώτα βήματα για να θεσμοθετήσουμε αυτή την ε, σχέση εργασίας με τον Ολυρέν και θα είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Ε, αυτό συνδέεται και με τις στρατηγικές εξόδου, εξόδου από την κρίση. Ε, πώς ε, τα διάφορα μέτρα υποστήριξης θα εξαλειφθούν βαθμιδών τα επόμενα χρόνια. Επομένως θα ήθελα να εστιάσω στην, ε, σε αυτά τα μέτρα και στην βαθμία κατάργησή του, σε συνδυασμό με την απασχόληση και να εξασφαλίσουμε ότι η έξοδος θα λάβει χώρα μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάκαμψη στις χώρες. Αυτό βέβαια εύκολο να το λέει κανείς, δύσκολο να το κάνει. Ε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχει συνεργασία με τον ομολογό μου. Τώρα για τα σχολεία και την κατάρτιση. Θα πρέπει να συνεργαστώ με την Επίτροπο κυρία Βασιλείου για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης. Θα πρέπει να συνεργαστώ με την ε, Επίτροπο κυρία Χίδεγκαρτ, Χάντεγκαρτ, συγγνώμη. Εξαρτάται από ποιο θέμα πιάνουμε. Πάντα θα πρέπει να έχουμε ομάδες εμπειρογνωμόνων όμως. Ε, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μια νέα ανακοίνωση, Φερρυπίν, για την προστασία του κλίματος. Και εργαζόμαστε για τις πράσινες θέσεις απασχόλησης υπάρχουν συγκεκριμένες παράγραφοι για αυτές τις θέσεις και γίνονται καλές συστάσεις στο κείμενο. Μπορούν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης πράσινες και πώς μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει, είναι τμήμα δηλαδή της ατζέντα μας. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι ό,τι αφορά τη μείωση της φτώχειας. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, μια συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, σε όλα τα κράτη-μέλη, όλων των διαφερομένων, ότι πραγματικά μπορούμε να θέσουμε στόχους μείωσης της στόχιας. Να συμφωνήσουμε γι' αυτό καταρχήν. Και αυτή τη στιγμή σε αυτό γίνει αποδεκτό, θα πρέπει να πείσουμε τους πάντες ότι μπορούμε να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με, το, με δεδομένο το χρονικό μας ορίζοντα. Έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να γίνει, αλλά μην ξεχνάτε την εξαιρετική δυσκολία κατά την αφετηρία. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι φέτος οι στατιστικές για την ανεργία θα είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικές. Ε, θα υπάρχουν επιπτώσεις ε, σε διάφορες χώρες για τα επόμενα χρόνια λόγω της κρίσης. Χωρίς όμως το στόχο αυτό μείωση της στόχιας, αποκλείεται τα κράτη-μέλη να ανασκουμποθούν και να ασχοληθούν με τα θύματα της κρίσης. Να ασχοληθούν με εκείνους που δεν έχουν ξαναβρει κάποια δουλειά και αποκλείεται να ασχοληθούν με εκείνους που έχουν χαμηλότατα εισοδήματα, που έχουν μεγάλες οικογένειες, που ζουν μόνοι τους και είναι γέροι και έχουν λίγα λεφτά παράλληλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο φετηρίας. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να ενδυναμώσουμε τα συστήματα κοινωνικής προστασίας, εκεί όπου είναι αδύναμα. Και θα συζητήσουμε με πολλές λεπτομέρειες ε, για αυτά τα θέματα στην κοινωνική ατζέντα. Θα είναι το επόμενο κείμενο μετά την, ε, τις κατευθυντήριες ε, για την εφαρμογή της ε, στρατηγικής ε, του 2020. Όταν αυτές ολοκληρωθούν, το επόμενο κείμενο, κοινωνική ατσέντα. Πάμε στον τρίτο γύρο ερωτήσεων, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Σιλβάνα Ράπτη είναι η πρώτη, Γιούτα Στάινμπεργκ μετά. Η κυρία Ράπτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τον Επίτροπο τον οποίο βλέπουμε συνεχώς με ευχαρίστηση στο Κοινοβούλιο. Ήταν στην ημερίδα που οργάνωσε ο κύριος Σέρκα, ήταν σε μια κοινή εκδήλωση με το ΣΕΝΤΕΦΟΠ και αυτό μας ευχαριστεί. Ωστόσο θέλω να ρωτήσω, άκουσα τους σχεδιασμούς για το 2020 και αναρωτιέμαι, έχουμε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει το 2010 γιατί ακούγοντας για το 2020 ε, νομίζω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακριβώς τι μας συμβαίνει στην Ευρώπη, στα κράτη-μέλη και συνολικά για το 10. Το πρόγραμμα Έρασμος για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Συμφωνώ, μου αρέσει. Όμως δεν γίνονται προσλήψεις. Άρα είναι ένα θέμα. Νέοι με προσόντα και γνώσεις. Μου αρέσει. Αλλά έχετε σκεφτεί, έχετε παρατηρήσει ότι νέοι που έχουν πολύ περισσότερα προσόντα πηγαίνουν σε δουλειές που δεν χρειάζονται αυτά τα προσόντα και παίρνουν λιγότερα χρήματα διαφορετικά δεν θα βρουν δουλειά. σκέπτομαι ότι καθώς βρίσκουμε διάφορους όρους που χρησιμοποιούμε μήπως πρέπει να βρούμε ακόμη έναν χειρονάκτες της γνώσης. το λέω στη γλώσσα μου δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. χειρονάκτες θα δουλέψω πάνω σε αυτό και θα σας κάνω πρόταση για αυτό τον καινούριο όρο, γιατί νομίζω ότι θα τον χρειαστούμε. Ε, απολυμένοι. Απολύονται άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Και στην α, ημερίδα που είχαμε με το Σεντεφόπ και ανταλλάξαμε και εκεί απόψεις, είπατε ότι θα πρέπει να συνεργαστείτε με την κυρία Βασιλείου, όπως το είπατε και εδώ. Ε, Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι αυτοί εκτός από επανεκπαίδευση έχουν και οικογένειες. Απομακρύνετε το κινητό σας. Ε, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι ε, σημαντικά προβλήματα και είναι προβλήματα της ζωής, σημερινά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, τελειώνω αμέσως, αμέσως, λέγοντας μία κουβέντα. Έχουμε μία παροιμία στην Ελλάδα που λέει το εξής. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι. Ελπίζω ότι η παροιμία αυτή δεν θα ισχύει για τη στρατηγική του 2020. Ευχαριστώ και έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά σας και στην προσπάθεια που θα κάνετε στην Επιτροπή. Euh, σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία και μετά η κυρία Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Ομολογώ ότι ε, θα περίμενα περισσότερα στο έγγραφο για την ποιοτική εργασία. Δεν μου φτάνει. Και θέλω να αντιδράσω σε αυτά που είπε ο κύριος Μαν. Δεν αρκεί να ακούς αυτά που λένε τα συνδικάτα, να συμπεριλαμβάνεις και καμία πρότασή τους καμιά φορά στα κείμενα. Πολλοί συνάδελφοι μίλησαν για τις επισφαλείς μορφές εργασίας. Ε, εγώ θα ήθελα να ε, ασχοληθούμε ε, με τους ε, φτωχούς εργαζομένους. Δεν είναι ότι είναι άνεργοι οι άνθρωποι, είναι ότι δουλεύουν, αλλά είναι φτωχοί στους χαμηλόμισθους. 14 εκατομμύρια στην Ευρώπη πλέον είναι εκείνοι που εργάζονται και είναι φτωχοί και ζουν κάτω από το κατόφλι της φτώχειας που είναι για τα ε, είδη πρώτης ανάγκης και το επόμενο διάστημα και τα επόμενα κατά την άποψή μου το έγγραφο δεν δίνει αρκετό χώρο σε αυτό αυτή την πραγματικότητα, γιατί και αυτό έχει σχέση με την κοινωνική ειρήνη στην Ευρώπη. Και άλλες στρατηγικές, πολύ συγκεκριμένε μου λείπουν εμένα από το εφό, Είπατε θα τα δείτε στη συνέχεια, αλλά μια παράκληση και εγώ, ιδιαίτερα ε, ευάλωτε ομάδε του πληθυσμού να αντιμετωπιστούν από ειδικέ στρατηγικέ και ε, χρειάζεται βοήθεια ε, για τους νέους, για τους μακροχρόνια άνεργους, για τους μετανάστες, για τις μονογονεϊκές οικογένειες κτλ. Η κυρία Κίνγκα Γκένς και μετά η κυρία Γκαμπρία Τσίμερ. Ε, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ε, παρέμβασή σας. Όλοι πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό το έγγραφο αυτό για τα επόμενα 10 χρόνια και γι' αυτό και αναζητούμε ε, να κατανοήσουμε τον περίπλοκο χαρακτήρα και αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι. Θέλω να κάνω κάποιες συστάσεις και ερωτήσεις. Οι συστάσεις αφορούνται, ε, εντάσσονται μάλλον στην ε, βελτίωση της ανάπτυξης. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της γύρανσης. Μιλάμε για την γυράσκουσα κοινωνία μας, αλλά πιστεύω πως ο γυράσκον πληθυσμός αποτελεί και πλονέκτημα για μας. Αν μπορούμε να τους συμπεριλάβουμε και να τους εμπλέξουμε περισσότερο, με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε στην αγορά εργασίας, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση βελτίωση της οικονομικής κατάστασης ε, αν έχουμε έναν υγιέστερο το πληθυσμό θα ήταν ίσως βοηθητικό και για το μέλλον. Να ε, το προτείνουμε αυτό ως ε, πλεονέκτημα. Τώρα για τον πληθυσμό το Ρώμα, ξέρω πως και εσείς είστε ιδιαίτερα προσιλωμένοι στο θέμα αυτό. Εχθές έγινε μια δημόσια ακρόαση και ακούστηκε μια πολύ ισχυρό αίτημα για την ανάπτυξη μιας ε, πανευρωπαϊκής στρατηγικής για τους Ρώμα. Ε, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει αν υπήρχε αρκετή διαθεσιμότητα στην πρόσβαση, στην κατάρτιση, στην παιδεία ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση για το μέλλον. Αναφέρονται και οι ανάπηροι, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες στο κείμενο. Αλλά νομίζω και εδώ θα χρειαστεί μεγαλύτερη υποστήριξη ώστε να συμμετέχουν περισσότερο. Και οι νέοι το ίδιο. Οι ερωτήσεις μου αφορούν περισσότερο την εφαρμογή. Αν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο θα εφαρμοστεί, νομίζω πως θα είναι πολύ σημαντικό. Πώς βλέπετε μια νέα προσέγγιση που να είναι από πάνω προς τα κάτω, να είναι πιο αποτελεσματική από την προηγούμενη της Λισαβόνας. Δηλαδή, αυτό από την μια πλευρά και από την άλλη πλευρά, πώς βλέπετε το μέλλον της πολιτικής συνοχής που είναι και πάλι πολύ σημαντικό για μας λόγω της πτυχής αλληλεγγύης για τη στρατηγική 2020. Ε, πώς το βλέπετε το μέλλον ε, σε σχέση με τη νέα προοπτική δημοσιονομικών προοπτικών για το 2014 και Επίσης, ποιος ήταν ο ρόλος των υφιστάμενων των πολιτικών στην εφαρμογή. Ευχαριστώ. Κυρία Τζίμερ. Λυπάμαι, κύριε Επίτροπε, αλλά κατά την άποψή μου από τη στρατηγική 2020 λείπει έστω και ένα ίχνος υποψία οράματος για την καταπολέμηση και την εκρίζωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εγώ θα ήλπιζα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα αντλούσε την έμπνευσή της και από τον ΟΗΕ και την εκεί συζήτηση που γίνεται. Και γιατί χρησιμοποιείτε τον ορισμό της σχετικής φτώχειας. Και για τους στόχους μιλάτε μόνο για 20 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν ε, σε συνθήκη φτώχεια. Και οι άλλοι τι γίνεται. Τι γίνεται με τους αστέγους. Φέτος το χειμώνα πέθαναν εκατοντάδες. Ειδικά στην Πολωνία πάνω από 220 άστεγοι. Δεν μπορούν όλα αυτά να ε, αποτελματωθούν στους, στα 20 εκατομμύρια των ανθρώπων που κινδυνεύουν να ζήσουν στη φτώχεια. Όλα αυτά είναι ένας χυλός, είναι ένας αριθμός που δεν μπορεί ούτε να μετρηθεί, ούτε να ελεγχθεί, ούτε να καταπολεμηθεί. Και από σαν τη Λισαβόνα που είχαμε μέχρι τώρα. Και μετά λέτε ότι η απασχόληση των γυναικών δήθεν αυξήθηκε και σημαντικά κιόλα. Σαν να μας λέτε ότι εντάξει, οι γυναίκες είναι ευτυχισμένες, δουλεύουν και τι φωνάζετε. Ναι, αλλά με ποιε συνθήκες και ποια κριτήρια δουλεύουν αυτές οι γυναίκες. Στη Γερμανία πάνω από 42% όλων των εργαζομένων γυναικών είναι σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στους άνδρες είναι 6,2% στη μερική απασχόληση. Αυτό το πουλάτε, το σερβίρετε ως επιτυχία. Εγώ θέλω να είμαστε εδώ πιο ειλικρινείς, πιο συγκεκριμένοι και να έχουμε και όραμα με στόχους πραγματικού που είναι η κατάργηση, η εκρίζωση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας στην Ένωση. Αυτό είναι το θέμα και όχι αυτή η γενική ε, ανακατοσούρα για να μπορεί να μην το ελέξει κανείς. Και σε πέντε χρόνια θα έρθετε να εξαγγέλλετε ότι τα 20 εκατομμύρια τα μειώσαμε. Εντάξει, και στον δρόμο θα είναι τα πάντα ίδια. Ο Επίτροπος. Οι στατιστικές είναι όντω ατελεί, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε την πρόοδο. Αυτό που είναι σημαντική αλλαγή είναι ότι η ικανότητα να διαμορφώσουμε μια καλή εικόνα για τις ε, κοινωνικές ε, συνθήκες και τις κοινωνικές σχέσεις, η εικόνα αυτή έχει βελτιωθεί. Γι' αυτό μπορούμε να θέσουμε στόχους και να μετρήσουμε την πρόοδο. Και αυτό ισχύει και για τους γενικούς οικονομικούς δείκτες, αλλά και για τους κοινωνικούς δείκτες. Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά και εμπιστοσύνη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κάθε κράτους μέλους ότι είμαστε σε θέση να καταλάβουμε πόσοι άνθρωποι κινδυνεύουν από τη φτώχεια και ποιες αλλαγές ε, συνέβησαν από δεκαετία σε δεκαετία. Φυσικά θα ήταν ιδανικό το να εξαλείψουμε μέσα σε 10 χρόνια τη φτώχεια. Θα ήταν ένα ιδανικό. Ε, θα ήταν ακόμα καλύτερο να την ε, εξαλείψουμε και σε ένα χρόνο μέσα. Ή και αύριο αν γίνεται. Ακόμα καλύτερα. Το θέμα είναι ρεαλιστικά τι μπορούμε να πούμε. Μέσα στο θεσμικό πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι μπορούμε να πούμε ρεαλιστικά. Συμφωνώ πλήρως ότι δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για τη στρατηγική τη δεκαετία αυτή, αλλά πρέπει να εστιάσουμε και σε το τι μπορούμε να κάνουμε. Μέσα στο 2010, μέσα αυτή τη χρονιά. Γιατί σήμερα ζούμε αυτή τη φοβερή κρίση ανεργίας. Και ίσως η βαθιά κοινωνική κρίση μας περιμένει τα επόμενα χρόνια. Δεν έχουμε, ένα, δεν έχουμε μια ιδανική λύση για αυτή την κρίση. Λείπει από τα βιβλία της οικονομίας, λείπει από τα βιβλία όλων μας, λείπει από την γνώση και από την εκπαίδευση που λάβαν οι εμπειρογνώμονες. Ακόμα και οι καλύτερες προβλέψεις δεν μας ε, οδήγησαν σε καλές αποφάσεις τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά πρέπει να τα δεχτούμε, να τα παραδεχτούμε και αποδεχτούμε. Αλλά νομίζω ότι το κείμενο για τη στρατηγική του 2020 μιλάει για την ανάγκη για οικονομικούς κανονισμούς και για ρυθμίσεις για να συνεχίσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα οικονομικής ανάκαμψης Και αυτό υπάρχει σε, εμποτισμένο σε μία πλειάδα πρωτοβουλειών. Αν κοιτάξετε το τίτλο για την απασχολησιμότητα, μιλάει και για ποσοτικούς στόχους, αλλά και για ποιοτικούς στόχους ε, σε ό,τι αφορά την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και επίσης, ε, εκεί που μιλάμε για την ε, βιομηχανική πολιτική στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, υπάρχουν εκεί σημαντικά σημεία για την εταιρική ευθύνη, φερρυπίν, αυτό το θέμα δεν πρέπει να το προωθήσουμε μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς. Ξέχασα στο προηγούμενο γύρο, απαντώντας, να αναφέρω το εξής. Έχουμε ένα σχέδιο να, να ασχοληθούμε με την γύρανση του πληθυσμού. Δεν θέλω να ανακατεύουμε τα εργαλεία, την, την ανεργία των νέων δηλαδή και πώς θα την αντιμετωπίζουμε και την ανεργία των γυρεότερων εργαζομένων. Νομίζω ότι θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε χωριστά. Θα πρέπει να δούμε τις συνθήκες απασχόλησης χωριστά των μεν και των δε. Και τις ευκαιρίες απασχόλησης που έχουν οι μεν και οι δε χωριστά. Και φυσικά να δούμε και, τις, και τα προβλήματα του γυράσκοντος πληθυσμού πρέπει να το δούμε πολύ περισσότερο γιατί οι δημογραφικές αλλαγές ε, τα τελευταία χρόνια έχουν επιταχυνθεί και θα αποτελέσει ε, σημείο εστίαση στην επόμενη περίοδο. Θα ξεκινήσουμε δραστηριότητες όπως η πράσινη βίβλος για τις συντάξει που θα εκπονηθεί ο νούπο. Αλλά αυτό είναι ένα σημείο αφετηρίας μόνο. Η κατάσταση των εργαζομένων και των συνταξιούχων άνω των 55. και θα ασχοληθούμε με τον ενεργό γυράσκοντα πληθυσμό ε, το 2012. Αυτά τα πράγματα, αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα λύσουμε μία νυχτή, αλλά ελπίζω με αυτή τη διαδικασία να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, το χαμένο χρόνο. Σίγουρα θα πρέπει να είχαν γίνει περισσότερα τα τελευταία χρόνια. Η δημογραφικές εξελίξεις ε, είχαν ήδη δημογραφικές επαναλαμβάνω εξελίξεις είχαν ήδη προβλεφθεί στη δεκαετία του 90. Τα ξέραμε όλα αυτά, αλλά τα, τα κράτη-μέλη μην ξεχνάτε ότι έχουν τη βασική ευθύνη για αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως θα πρέπει να συνεργαστούμε για να για τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, πολιτικές συνοχής. Τι σχέση υπάρχει μεταξύ της στρατηγικής του 2020 και τα μέσα για τη συνοχή, τα εργαλεία για τη συνοχή. Ακούστηκε ένα σχόλιο ότι τη συνοχή δεν θα πρέπει να τη βλέπουμε ως μια δέσμη εργαλείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ως ένα αυτόνομο στόχο. Έτσι θα την αντιμετωπίσουμε και θα συζητήσουμε πολύ περισσότερο το θέμα της συνοχής ε, κατά την αναθεώρηση τη δημοσιονομική. Α, ναι, και η Ρώμα. Στον προηγούμενο γύρο εξήγησα ήδη πώς βλέπουμε την συνέχεια που θα δοθεί στους στόχους ε, για την καταπολέμηση της στόχιας. Καλό παράδειγμα είναι αυτό που δώσατε. Θα πρέπει απλώς να περιμένουμε τη μείωση της στόχιας μόνο και μόνο επειδή κάποια στιγμή θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη και θα δημιουργηθούν θέσει απασχόλησης γενικά. Υπάρχουν διάφορες ομάδες, συγκεκριμένε ομάδες που είναι περιθωριοποιημένες και υπάρχουν λόγοι που δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας, στις δικές τους χώρες. Γι' αυτό λοιπόν θα ενδυναμώσουμε τις πολιτικές για τους Ρώμα. θα υπάρξει μια νέα ανακοίνωση από την κυρία Ρέντιν και από μένα που θα εκδοθεί αυτό το μήνα, στο τέλος του Μαρτίου. Και θα πάμε μαζί τον Απρίλιο στην ε, Σύνοδο για τους Ρώμα, στην Κόρδοβα. Και εκεί θα μιλήσουμε για τις ενισχυμένες πολιτικές κομισιών για τους Ρώμα, στη Σύνοδο αυτή της Κόρδοβας. Πάμε Ευχαριστώ. Περνάμε στο τέταρτο γύρο ερωτήσεων και η πρώτη από αυτές θα τεθεί από την κυρία Εβελίν Ρενιέ και μετά η κυρία Ελιζαμπέτ Σρέντερ. Τρεις ερωτήσεις κύριε Επίτροπε έχω, αλλά προηγουμένως θα ήθελα να σας συγχαρώ ειλικρινά για ε, τα όσα είπατε απέναντι στον αυστριακό τύπο για το ρόλο των τραπεζών της χώρας, της χώρας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Πάνει, έχω διαβάσει τόσο σαφή και στερά τα λόγια. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ρόλος των νέων ηλικίας 15 έως 20 ετών. Το λεγόμενο διτό σύστημα εκπαίδευσης με ε, σχολείο και μαθητεία είναι πολύ σημαντικό και μπορεί να είναι πολύτιμο για την αγορά εργασία και το έγγραφο δεν με ικανοποιεί γιατί αρχίζει στην ηλικία των 20 ετών. Ερώτηση δεύτερη. Η φτώχεια και η καταπολέμηση της πολλά υπόθηκαν ήδη σχετικά. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω κι εγώ κάτι. Παρακαλώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια στάση έχει και πώς φαντάζεται την καταπολέμηση της φτώχειας ε, όταν στο ε, κείμενό τη λέει τόσα λίγα για τις κοινοφελεί υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι δημόσιες κοινοφελείς υπηρεσίες για την συνοχή της κοινωνίας. Και φαντάζομαι ε, ότι είναι σημαντικός ο ρόλος εκεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα πρέπει κάτι να πείτε. Και η τρίτη ερώτηση αφορά ε, το μέλλον των κοινωνικών ελαχίστων προδιαγραφών από όλα αυτά που μας είπατε δεν έχω καταλάβει ακόμα πώς συγκεκριμένα φαντάζεστε το μέλλον των ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών. Γιατί όλα αυτά είναι πιο μακρινά, πιο εξωτικά και πιο απόμακρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρωτοβουλίες για τις αναδιαρθρώσεις, ας πούμε, ε, για το ωράριο εργασίας για τις αποσπάσεις εργαζομένων. Είναι τεράστιο πεδίο. Και επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα και τα είπαν πολλοί προλαλήσαντες ε, και προλαλήσασες, πάρα πολύ σημαντικό μέσο, θα ήθελα τη γνώμη σας. Η κυρία Και μετά η κυρία Ραγκίνα Μπάστος. Ευχαριστώ. Κύριε Επιτροπέ, θα ήθελα να επανέλθω σε δύο σημεία που αναφέρθηκαν και προηγουμένως και η απάντησή σας ε, δεν με κάλυψε. Πρώτον, οι πράσινες θέσεις απασχόλησης είναι απορίας άξιος. Παρά τη δημόσια συζήτηση που γίνεται για το θέμα, παρά τις προεργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πού είναι η οριζόντια γραμμή, η εγκάρσια γραμμή στο 2020, πουθενά δεν φέρεται αυτός ο Ιρμός ε, στη σκέψη σας. Δηλαδή, ε, εντάξει η πράσινη οικονομία, εντάξει η έξυπνη οικονομία, που συνδέεται αυτή με την απασχόληση. Κάποιος συνάδελφος το ανέφερε αυτό ήδη, γιατί υπάρχουν θέματα πάρα πολύ ευαίσθητα τι ποιότητα θα έχουν οι αίσθησεις απασχόλησης, ποιες θα είναι οι βασικές προδιαγραφές και τα στάνταρ, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι νέες θέσεις απασχόλησης να είναι χειρότερες από τις προηγούμενες και αυτό δεν το λαμβάνεται υπόψη. Και το δεύτερο βασικό θέμα που με απασχολεί είναι ακριβώς η μετάβαση από τη σημερινή οικονομία στην επόμενη. Σήμερα η κατάσταση πώς έχει, και αυτό το βλέπουμε και σε πολλές μελέτες ε, οργανισμών και αρμοδίων. Χάνονται θέσει απασχόληση, δημιουργούνται νέε. Εμεί πώ το αντιμετωπίζουμε αυτό, Πώ αντιμετωπίζουμε τον κόσμο που αγωνιά με χάσει τη δουλειά του, Ποια είναι η ευθύνη μα και πώ την αναλαμβάνουμε, Και εμεί και οι επιχειρήσει όμω για την κατάρτιση, τη μετεκπαίδευση των εργαζομένων και αυτή η κοινωνική εξασφάλιση στη μεταβατική αυτή διαδικασία, στο μετασχηματισμό προς τη νέα την πράσινη οικονομία, πώς συνοδεύεται. Ε, ε, εκεί είναι οι εγκάρσιες συνδέσεις που προσφέρεται ακριβώς η στρατηγική 2020 για αυτή. Τίποτα δεν βλέπω σχετικά, δεν με ικανοποιεί το έγγραφο. Θα δεν... Και δεν με ικανοποιεί και η απάντηση θα εκδώσουμε ανακοίνωση. Όχι. Να μας πείτε από σήμερα ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι σας στόχοι έστω και αν τους φέρετε αργότερα με μορφή νομοθεσίας ή διαδικασίας, τουλάχιστον οι στόχοι σας ποιοι είναι συγκεκριμένα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπάστος και μετά ο κύριος Κρίστενσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τον Επίτροπο και ευχαριστώντας ε, την, τον για τον διάφανο τρόπο με τον οποίο έκανε την παρέμβασή του, την παρουσίασή του, αλλά και τις απαντήσεις του και κυρίως για τη ρεαλισμό του σε σχέση με την κρίση που διανύουμε και το ότι δεν έχει φτάσει στην αρνητική ε, κορύφωσή της, τουλάχιστον σε θέματα απασχόλησης. Αυτή η στρατηγική 2020 θεωρούμε πως δεν είναι μόνο μια στρατηγική για την επόμενη δεκαετία, αλλά είναι μια πολιτική πιο μακροπρόθεσμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μπορέσει να συγκεκριμενοποιήσει μια δίκαιη και ίση κοινωνικο-οικονομική πολιτική για ε, το μέλλον. Η πρώτη λοιπόν πρωτοβουλία είναι η απάντηση στην κρίση και η φιλοδοξία ο κόσμος να μπορέσει να επανέλθει στην αγορά εργασίας. Σε σχέση με αυτό το θέμα, εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε ένα θέμα το οποίο ήδη αναφέρθηκε εδώ και το οποίο ανέφερε και ο Επίτροπος και έχει να κάνει με την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Ο Επίτροπος μίλησε στο πλαίσιο της δράσης για την διευκόλυνση της εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας και ως προς αυτό μιλήσατε για την δημιουργία ενός μέτρου για το έρασμος πρώτη απασχόληση. Καταρχήν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα πέρα από αυτό το έρασμος πρώτη απασχόληση που αναφέρατε. Αναφέρεται ένα αντιφατικό στόχο, καταρχήν παραμονή, ε, έρχεται μάλλον σε αντίφαση με την παραμονή των πιο ηλικιωμένων στην αγορά εργασία. Είναι ένα στόχο τον οποίο επιδιώκουμε εδώ και καιρό. Ξέρουμε πω η Ευρώπη έχει πολύ σοβαρά δημογραφικά προβλήματα, ότι το προσδόκιμο ζωή είναι πολύ ψηλό, το οποίο είναι θετικό, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν κοινωνικά προβλήματα και ασκείται και τεράστια οικονομική πίεση στα δημοσιονομικά των κρατών μελών λόγω του προβλήματος του δημογραφικού. Άρα λοιπόν πώς εσείς συνδέετε την παραμονή των πιο ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας, πώς προωθείτε τους, την δραστήρια, την ενεργή γύραση και ποια είναι τα μέτρα που προτείνετε Ε, μέσα στο πλαίσιο αυτής της μεταρρύθμισης. Άλλη ερώτηση έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλήσατε παρόδο για τις μικρομεσαίες. Για μας Επιτροπή Απασχόλησης οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ένα ζωτικό μέσο, ένα εργαλείο για τη δημιουργία των νέων θέσεων απασχόλησης και για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης που αποτελούν το κινητήρα της δημιουργίας των θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα ήθελα να γνωρίζω αν έχετε κάποιο καινοτόμο και συγκεκριμένο μέτρο σε σχέση με τις πολιτικές για τις ΜΜΕ. Και τέλος, σε σχέση με τα όσα είπατε για τον ανοιχτό συντονισμό. Ξέρουμε πως τα κοινωνικά μέτρα και η κοινωνική πολιτική εμπίπτουν στην αρμοδιότητες των κρατών μελών και ότι πιθανότατα η στρατηγική της Λισαβόνας αν και όλοι μας θα πρέπει να αποκομίσουμε τα απαραίτητα δείγματα, δεν λειτουργήσε ακριβώς γιατί δεν υπήρξε ε, σοβαρή δέσμευση από πλευρά των κρατών μελών στην εφαρμογή της και στην συγκεκριμένη των στόχων που είχαν καθοριστεί από αυτή τη στρατηγική. Ένα από τα μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν για να μπορέσουν ε, τα κράτη να αναπτύξουν και να θυλοποιήσουν τις ε, τους στόχους της στρατηγικής ήταν ο μέθοδος τη ανοιχτού συντονισμού, που όπως γνωρίζουμε δεν είχε ιδιαίτερα εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μήπως λοιπόν ε, αυτός ο συντονισμός θα μπορούσε να γίνει έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να δεσμευτούν σε κοινωνικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν και η στρατηγική 2020 να έχει καλύτερη έκβαση από τη στρατηγική της Λισαβόνας έτσι. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Όλε Κρίστενσεν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εντάξει, υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία στη στρατηγική 2020, αλλά το θέμα είναι αρκετά φιλόδοξα. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Γίνεται λόγος για δύο διαφορετικά μέσα, δύο διαφορετικά εργαλεία στο έγγραφο. Το ένα είναι ε, η περιστολή ε, των δημοσίων λιμάτων ε, από τη μια και από την άλλη η ίδια η στρατηγική για το 2020. Εμένα με τρομάζει λίγο αυτό. Γιατί ε, αυτά τα χρηματοπιστωτικά θέματα του παρόντος μπορούν να επηρεάσουν ε, την εξέλιξη ε, για το μέλλον. Μέχρι το 2020 να μην προλάβουμε να δημιουργήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. δύο λόγος γίνεται στην έκθεση επίσης στο έγγραφό σας για το κοινωνικό dumping η κυβέρνησή μας και η Βουλή της Δανίας έχουν ήδη αντιδράσει, έχουν δώσει τα σχόλιά τους για το κείμενο αυτό 2020 ε, και ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει βήματα για να καταπολεμήσει το κοινωνικό ε, dumping. Σε πολλές χώρες υπάρχει πρόβλημα με τους λεγόμενους ψευδοαυτοαπασχολούμενους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βάλει κριτήρια. Τι εστί αυτοαπασχολούμενος, ποιος είναι ο ελεύθερος επαγγελματίας και πώς αυτό ε, στρεβλώνει ε, τον ανταγωνισμό στην Ευρώπη. Στη Δανία κάθε χρόνο έχουμε ε, μεγάλο αριθμό εργαζομένων, εκατομμύρια ολόκληρα που περνούν τα σύνορα και εργάζονται στη Γερμανία. Ε, ψεύδο αυτό απασχολούμενοι ε, και κερδίζουν 3 με 4 ευρώ την ώρα με πολύ επισφαλείς συνθήκε ε, και καταστάσεις. Αυτό είναι κοινωνικό ντάμπινγκ και πρέπει να καταπολεμηθεί. Ευχαριστώ. Uh, too much fiscal consolidation. Uh, Περιβολικά πολύ φορολογική παγίωση. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε, κυρίως την πρώιμη Μιλάμε για μια στρατηγική τη στιγμή που σε ορισμένα κάτι μέλη οι χρηματοπιστωτικέ αγορέ είναι αυτέ που καθορίζουν τα μέτρα για την έξοδο. Το θέμα λοιπόν είναι να, να ανακτήσουμε τον έλεγχο του τι συμβαίνει και το πώ οι φορολογικέ πολιτικέ ε, ε, ασκούνται και μετά να λάβουμε υπόψη ευρύτερα τις επιπτώσεις στην απασχόληση και στην κοινωνική πολιτική. Αλλά δεν νομίζω πως τονίζεται υπερβολικά. Επίσης θα πρέπει να δούμε πως ε, Όντως ε, τα θέματα αυτά θα είναι διαρκώς στην ημερήσια διάταξη τα επόμενα χρόνια και αναπόφευκτα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων στα κρατημέλη. Το ζήτημα είναι να έχουμε σχεδιάσει μια βάση ώστε να το εφαρμόσουμε με σεβασμό στους στόχους. Και βέβαια να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που θέτουμε μέσω της στρατηγικής 2020. Είναι δύσκολο να αναπτύξει κανείς περισσότερο την υπόθεση της κοινωνικής, του κοινωνικού dumping. Θα έλεγα ότι οι συνέπειες της άνεσης ανάπτυξης, του άνεσου επίπεδου εισοδημάτων στα κράτη-μέλη, οδηγούν σε αυτό. Και πάλι και εκεί πολλά μπορούν να γίνουν σε αυτό το τομέα, συμφωνώ. Ίσως θα έπρεπε να αναμένουμε περισσότερο από την κοινωνική ατζέντα σε σχέση με το συγκεκριμένο κείμενο και βέβαια στους διάφορους, ε, στα διάφορα θέματα όπου αντιμετωπίζονται οι συνέπειες του άνισου επίπεδου εισοδημάτων και εξελίξεων όπως για παράδειγμα η όθηση των εργαζομένων. σε σχέση με το ρόλο των... της ε, καινοτομίας και της ε, δημιουργίας των επιχειρήσεων. Αυτό έχει αναγνωριστεί από όλους τους επιτρόπους στη συζήτηση. Δυνατότητες δηλαδή για στήριξη μέτρων ξεκινώντας από την μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου, την ε, μικροχρηματοδότηση, την τροποποίηση των ε, συστημάτων κτλ. Δεν είναι μόνο μία η λύση για να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια ολόκληρη σειρά εργαλείων που θα τους βοηθήσουν να μπουν σε μια θετική πορεία. Ηλικία συνταξιοδότησης. Και πρότασή μας είναι σε σχέση με τους ηλικιωμένους που είναι ενεργεία στην αγορά και στην αγορά εργασίας. Τώρα εγώ δεν κρατώ κάποια συγκεκριμένη θέση σε διεθνή πλαίσια, αλλά θα πρέπει νομίζω να δούμε ήδη πριν φτάσουμε στα συμπεράσματα των συζητήσεων για την δραστήρια γύρανση και και το θέμα των συντάξεων πριν να φτάσουμε σε συμπεράσματα που είναι εύκολο να δει κανεί πως υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση που μπορούμε να ακολουθήσουμε στη μεταρρύθμιση των ορίων ε, συνταξιδότηση, να το αυξήσουμε δηλαδή όχι μόνο σου είναι επέος της κρίσης εγώ δεν θέλω να το βλέπω ως ε, ένα μέτρο που απλά εξηγείται μέσα στο πλαίσιο μιας κρίσης αλλά κυρίως πρόκειται για μια συνέπεια των δημογραφικών αλλαγών και έτσι θα πρέπει να το δούμε ρεαλιστικά όπως υπογραμμίστηκε και από κάποιον από τους ομιλητές. Για τους νέους έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για τη πρώτη ε, απασχόληση. Αυτή ήταν η ερώτηση νομίζω. Αυτό αναπτύσσεται φέτος ε, το πρόγραμμα και ε, αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί του χρόνου. Βελτίωση τη αντιστοιχία ανάμεσα στι θέσει επασχόληση και τι ανάγκε των ζητούντων εργασία. Αυτό είναι το, χρονοδιάγραμμα το οποίο δουλεύουμε. Δεν είναι κάτι που ε, αφορά το απότερο μέλλον, αν και θα πρέπει να σας ομολογήσω θα... θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουμε την ε, σοβούσα κρίση. Για τις δημόσιες υπηρεσίες υπάρχει ήδη δουλειά. Θα πρέπει να κατανοήσετε πως πρόκειται για ένα άγραφο με περιορισμένο αριθμό σελίδων και σειρών. Αλλά γίνεται ήδη σχετική συζήτηση με τον συνάδελφο Μπαρνιέ. Ήδη ξεκινήσαμε ανταλλαγή απόψεων. Και ε, θα επανέλθουμε. Ίσως να μην ε, αναφέρετε παρκώς ή όσο θα θέλατε. Αλλά η δουλειά συνεχίζεται και θα έρθουμε για να το συζητήσουμε και μαζί σας. Τώρα και πάλι για τους νέους τι πιστεύουμε για τις ηλικιακές ομάδες ανάμεσα στα 15 και τα 20. Γι' αυτό ακριβώς έχει μετακινηθεί ο... το πεδίο μάλλον στόχου για να δείξουμε ότι μάθαμε από τη Λισαβόνα και πρέπει να τονίσουμε για τους νέους την παιδεία σε αντίθεση με την ε, γρήγορη μετάβαση από τα σχολεία στην αγορά εργασίας. Είναι πιο ρεαλιστικό να θεσπίζουμε Υψηλού στόχους απασχόλησης για τις ομάδες τις ηλικιακή από τα 20 μέχρι τα 65 και να δούμε πώς η παιδεία, η κατάρτιση και η πρώτη εισαγωγή στην αγορά εργασίας των νέων θα μπορούσε να βελτιωθεί. Είναι κάτι αυτό που θα πρέπει λοιπόν να το στοχεύσουμε και να μειώσουμε και τα περιστατικά όπου τα παιδιά σταματούν το σχολείο. DOMC. Ε, we can have, ε, again and again Η ε, ανοιχτή μέθοδος συντονισμού είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως. Πώς να ενισχυθεί, πώς να βελτιωθεί Νομίζω θα πρέπει να επανέλθουμε ε, όταν θα είμαστε στις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή όλων αυτών των προτάσεων. Ευχαριστώ. Φτάνουμε στην τελευταία ομάδα ερωτήσεων. Η κυρία Παπαδοπούλου και εν συνεχεία ο κύριος Τόμας Χάντελ. Κυρία Ανιγόνη Παπαδοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή συνεδρία. Η ερώτηση μου είναι ξεκάθαρη. Εάν δούμε γύρω μας υπάρχει γενιά των νέων επιστημόνων των 700 ευρώ. Υπάρχουν οικογένειες που με 1000 ευρώ πρέπει να τα φέρουν βόλτα στο σπίτι. Υπάρχει η περιθωριοποιημένη τάξη των ηλικιωμένων εργαζομένων. Οι μονογονεί, οι μετανάστες, οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Τα άτομα με αναπηρία δεν νομίζετε ότι θα μπορούσε να ήταν πιο εξειδικευμένε και στοχευμένε οι στρατηγικέ ώστε για αυτέ συγκεκριμένα τι ομάδε να έχουμε πιο απτά αποτελέσματα. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη, όσον αφορά τους στόχους της στρατηγικής του ΕΕ2020, θεωρώ ότι είναι πολύ φιλόδοξη. Φαίνεται να είναι θεωρητικά πιο απλή και εστιασμένη, αλλά προϋποθέτουν πλήρη ανάκαμψη από την κρίση όλων των χωρών μελών και μετά ενα ένα νέο κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Με δεδομένο ότι η κρίση έχει χτυπήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικών τρόπων και η ανάκαμψη ποικίλει από χώρα σε χώρα και αντιμετωπίζονται πολλά εθνικά προβλήματα. Πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτοί οι φιλόδοξοι στόχοι της στρατηγικής θα υλοποιηθούν ομοιόμορφα με την ίδια ταχύτητα στα επόμενα δέκα χρόνια από όλε τι χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξεκινούμε με πολύ ανομοιόμορφη κατάσταση. Και η τελευταία με ερώτηση αφορά το εξή. Επειδή δεν μου αρέσει να μιλούμε μόνο θεωρία και πρέπει πρακτικά να δούμε πώ εφαρμόζεται η στρατηγική, χρειάζεται πρώτον και κύριον η πολιτική βούληση όλων των χωρών μελών. Υπάρχει. Χρειάζονται ρεαλιστικέ στρατηγικέ και κοινοτικό συντονισμό. Υπάρχουν. Χρειάζεται μηχανισμό παρακολούθηση τη υλοποίηση τη στρατηγική του 2020. Υπάρχει αυτό ο μηχανισμό. Είναι ξεκάθαρο. Χρειάζονται διορθωτικέ παρεμβατικέ ενέργειε. Ποιο θα τι κάνει αυτέ τι ενέργειε. Και τελευταία, χρειάζονται δείχτε σύγκριση των επιδόσεων κάθε χώρα όσον αφορά την επίτευξη των στόχων και αξιολόγηση ακριβώ τη συλλογική κοινωνική προσπάθεια. Υπάρχουν τέτοιοι ποσοτικοί και μετρήσιμοι δείχτες ώστε να δούμε και έμπρακτη εφαρμογή. Η εμπειρία που είχαμε μέχρι σήμερα για την καταπολέμηση της ανισότητας στα φύλλα, της καταπολέμηση ε, καταπολέμησης της φτώχειας, της εξέλιξης με τους στόχου της χιλιετίας του Οργανισμού είναι τέτοιες που δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι τι μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 τούτη τη φορά δεν θα μείνει στα λόγια αλλά θα υλοποιηθεί στην πράξη. Α, εξεπλάγει. Δεν περίμενα να πάρω το λόγο, κυρία Πρόεδρε. Α, να ανάβατε και κανένα μικρόφωνο, θα σας άκουγε και ο μιλητής που του δίνετε το λόγο. Ε, πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω τι γίνεται στη Γερμανία όταν ακούμε τέτοιες συζητήσεις. Μια τρύπα στο νερό θεωρούν στη Γερμανία ότι προσπαθείτε να κάνετε. Λίγα ήταν τα συγκεκριμένα και μέχρι τώρα αυτά μας τα λέγανε και ο Σπίτλα και ο Μπαρόζο αυτά που μας είπατε εσείς. Δεύτερο, αυτή η στρατηγική για το 2020 που έχουμε μέχρι σήμερα είναι μια διαδικασία από πάνω προς τα κάτω. Δεν συμμετέχουν ε, οι ενδιαφερόμενοι. Δεν ενδιαφέρεστε το καν να δώσετε την εντύπωση ότι οργανώνεται ένα στοιχειώδη δημόσιο κοινωνικό διάλογο. Γι' αυτό ε, ακούμε και επικρίσεις από πολλά συνδικάτα από την Ευρώπη, από πολλές κοινωνικές ομάδες, ότι για να αναπτυχθεί μια τέτοια στρατηγική πρέπει να αναλύσουμε λογικά τη στρατηγική της Λισαβόνας και τα αποτελέσματά της και όχι τώρα ε, στο γόνατο να κάνουμε νέες προτάσεις. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις, ίσως να μπορούσατε να τις απαντήσετε και εσείς ε, συγκεκριμένα. 60% επισφαλής θέσης εργασίας έχουμε στη δύση της Λισαβόνας. Πολύ φλέξη έχουμε και λίγο security. Κύριε Επίτροπε, δεν μπορεί κανείς να σας αποσπάσει αυτή τη δήλωση ότι να φτιάξουμε δουλειά και θέσεις απασχόλησης για να μπορεί να ζει από αυτές ο κόσμος χωρίς επιπλέον επιδόματα. Μπορείτε να το ξεστομίσετε αυτό το πράγμα. Δεύτερη ερώτηση. Ε, ε, η κοινωνική εταίροι θα πρέπει ε, να ενισχυθούν ε, στις δυνατότητές τους. Ναι, τι είναι αυτό, τι θα πει αυτό. Αυτό ουδέτερα ωραία λόγια είναι κενά. Ούτε ε, συνδικάτα ε, συμμετέχουν και υπάρχουν ακόμα εχθρικές προς τα συνδικάτα και τις συλλογικές συμβάσεις αποφάσεις του ΔΕΚ. Και λέει και ο Μπαρόσο δηλώνει ότι δεν θα αφήσει να θυγούν ε, ε, δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα της απεργίας και κάποια άλλα βασικά για το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Ερωτώ, πώς θέλετε να αλλάξετε το θεσμικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο για να ανταποκριθείτε σε αυτή τη δήλωση. Euh, Ευχαριστώ κύριος Λούτβιξον και μετά κύριος Δερόσα. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σας βλέπω μεταξύ μας. Ε, κύριε Επίτροπε, ελπίζω να σας δεχτούμε πολλές φορές και να ανταλλάξουμε απόψεις για να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό διάλογο, γιατί μόνο με στο διάλογο παίρνουμε καλέ αποφάσει. Προσπάθησα να συγκρίνω τη στρατηγική τη Λισαβόνα με αυτή την ε, στρατηγική του 2020. Και όντω υπάρχουν ε, λιγότεροι στόχοι σε αυτή τη νέα στρατηγική. Αυτοί οι στόχοι ε, είναι πιο εύκολα προσμετρήσιμοι. Το 2020 ίσως μας φαίνεται μακρινό, αλλά ξέρετε, ο καιρός περνά πολύ γρήγορα. Και ξέρουμε ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Τώρα, πώς θα τα καταφέρουμε ούτω ώστε να προχωρήσουμε με γοργό βήμα. Πώς θα τα καταφέρουμε αυτή η στρατηγική του 2020 από τη στιγμή της υιοθέτησής της να μην μείνει μέσα στα σιρτάρια. Αυτό το κείμενο θα πρέπει πραγματικά να επικαιροποιείται, θα πρέπει να το έχουμε μπροστά στα μάτια μας συνέχεια, θα πρέπει συνέχεια να επαληθεύουμε ότι προχωράμε καλά, ότι γίνεται σεβαστό, θα πρέπει να κάνουμε εκθέσεις στην Επιτροπή, να κάνετε στην Επιτροπή απασχόληση και στο Κοινοβούλιο Γέννη για τον τρόπο με τον οποίο η στρατηγική του 2020 λειτουργεί και, με τον τρόπο με τον οποίο, και για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι στόχοι. Εγώ συμμερίζομαι πολλέ από τι κριτικέ του κυρίου Σέρκα. Δεν θα τι επαναλάβω λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Αυτό είναι εκ των ονουκάνευ. Πρέπει να αποφύγουμε να φτάσει το 2020 και να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν κάναμε αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Το να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ένα το κρατούμενο. Αλλά το να μην κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Και σας ευχαριστώ που μας αφιερώνετε το χρόνο σας και απαντάτε στις ερωτήσεις. Έχω πολλές ερωτήσεις. Και καθώς ε, ε, ακούγονται περισσότερες παρεμβάσεις, ε, μεγαλώνουν οι ερωτήσεις μου. Για τις κοινωνικές υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος, θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα. ποια είναι η προσέγγισή σας στην ιδέα μιας οδηγίας για τις κοινωνικές υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος. Ε, χάρηκα που μιλήσατε στον Επίτροπο Μπαρνιέ για το θέμα αυτών των ε, υπηρεσιών, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Φαντάζομαι ότι έχετε ένα θεμελιώδη ρόλο που μπορείτε να παίξετε σε αυτόν τον τομέα. αναφέρθηκε ήδη το θέμα της στόχιας στην Ευρώπη. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν περίπου 85 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών που ζουν είτε μέσα στη φτώχεια είτε κινδυνεύουν. Αυτή είναι απαράδεκτη κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να την ε, ξεπετάξουμε έτσι εύκολα και να πούμε «Α, ελπίζουμε ότι η οικονομική ανάπτυξη θα βγάλει κάποιους ανθρώπους από τη φτώχεια ή θα τους εμποδίσει να πέσουν κάτω από το όριο». Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι η πρόσβαση στις κοινωνικές ε, υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος είναι βασικό στοιχείο για να εξασφαλίσουμε ότι ο κόσμος μπορεί να και είναι σε θέση να αποφύγει τη φτώχεια ή να, να ελαφρύνουμε το άχθος για αυτούς που ζουν σε συνθήκες ένδυας. Οι κοινωνικές λοιπόν υπηρεσίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το θέμα αυτό. προσπελασιμότητα, ε, καλές τιμές και υψηλή ποιότητα. Η συνθήκη της Λισαβόνας μιλάει για αυτό το θέμα σε ένα νέο άρθρο και σε ένα νέο πρωτόκολλο και ελπίζω ότι θα βρείτε έναν τρόπο ούτω ώστε να δημιουργήσετε και ένα νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές κοινωνικέ υπηρεσίες και να το βασίσετε σε αυτές τις νέες διατάξεις αγώνα. Τώρα για ένα πιο γενικό θέμα τη ε, κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Θα ήθελα να πω ότι ο Τιτανικός ε, βυθίστηκε όχι γιατί ήταν ένα κακό από μηχανική άποψη ε, πλοίο, αλλά γιατί προσέκρουσε ε, σε ένα παγόβουνο κάτω από, το, την επιφάνεια της θάλασσας. Δεν ήταν προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο. Σήμερα χτίζουμε, φτιάχνουμε πλοία για να και εξασφαλίζουμε ότι δεν θα βυθιστούν για τον ίδιο λόγο αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε μάθει τα μάθημά μα. Διότι αφωνώ μαζί σα ότι τα βιβλία, ας πούμε, δεν μα έχουν μάθει να αντιμετωπίζουμε τι καταστάσει που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιε κρίσει, κοινωνικέ κρίσει, τουλάχιστον από τι αρχέ τη δεκαετία του 90 σε διάφορε περιοχέ του κόσμου, όπου τα οικονομικά συστήματα. Ε, μην ανυπομονείτε, θα, θα, θα κλείσω όπου να είναι. Ε, τα χρηματοπιστωτικά συστήματα γονάτισαν τι οικονομίε να μην ξεχνάμε ότι οι υπερφιλελεύθερες πολιτικές θα μας ξαναβουλιάξουν αν δεν αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, χειραγώγησης των ε, ε, χρηματαγορών. Δεν μπορούν αυτές να μας εξουσιάζουν. Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να τις ελέγξουμε αυτές τις αγορές. Να ξεκινήσω από το τέλος, λέει ο Επίτροπος. Έχουμε παρόμοιες απόψεις για τις, τα αίτια της κρίσης. Και ακριβώς γι' αυτός, γι αυτό το λόγο ε, υποστηρίζω ανεπιφύλακτα τον Επίτροπο Μπάγνια για τις, ε, την προσπάθειά του να ρυθμίσει τις αγορές. Επίσης, συμφωνώ ότι θα πρέπει την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας να την διορθώσουμε μέσα από την διόρθωση της ατζέντα μας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι λείπουν αυτά τα πράγματα που ζούμε σήμερα από τα βιβλία. Είναι άνευ προηγουμένου η κρίση, είναι τέτοια η πτώση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στη μεταπολεμική περίοδο. Το μόνο συγκρίσιμο στοιχείο είναι το μεγάλο κράχ του 29, στη δεκαετία του 30, όπου δεν υπήρχε τότε δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και βλέπετε ότι η Κομισιόν ε, πολύ γρήγορα εκπώνησε ένα κείμενο με την ε, ιδέα πούμε, στο μυαλό τη, ότι σε μια τέτοια κατάσταση χρειάζεται ένα έντυπο. Ίσως δεν έχει όλες τις λεπτομέρειες, δεν έχει όλες τις απαντήσεις, αλλά δημιουργεί ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να προδεύσουμε. Πώς θα προδεύσουμε τώρα ταχαίως ήταν ένα από τα ερωτήματα που θέσατε. Το πιο σημαντικό νομίζω είναι να συμφωνεί στο Συμβούλιο και να αντιπαρατεθούμε στις απόψεις ότι η φτώχεια θα εξαλειφθεί απλά και μόνο με την αύξηση της απασχόλησης σε μια μεταγενέστερη φάση και να αντιταχθούμε στις απόψεις ότι η επιχειρηματικότητα από μόνη της θα εντείνει την απασχόληση χωρίς κυβερνητικές προσπάθειες και χωρίς συντονισμένες κυβερνητικές προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ πλήρως ότι ο στόχος της στόχιας είναι κρίσιμος και οι κοινωνικές υπηρεσίες καθολικού ενδιαφέροντος επίσης θα παίξουν κεφαλαιόδη ρόλο στην αντιμετώπιση της στόχιας. Τώρα, το αν θα υπάρξει οδηγία γι' αυτό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις τεράστιες διαφορές στα κράτη-μέλη και την, α, τις διαφορές και ποικιλομορφίες που σας παρουσίασα στην αρχή της α, παρέμβασής μου. Το έχω συζητήσει αυτό και σε προηγούμενες επαφές με την Επιτροπή και αυτό που ετοιμάζουμε είναι ένα ποιοτικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς αυτά τα θέματα που είπατε, την πρόσβαση, την ποιότητα ε, και τις προσιτές τιμές. Εν συνεχεία, λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μετά την εκπόνηση αυτού του πλαισίου. Τώρα, κάτι ενδιαφέρον. Άκουσα ότι αυτή η στρατηγική ήταν φιλόδοξη. Είπατε βεβαίω ότι θα πρέπει να είχαμε θέσει ακόμα πιο φιλόδοξου ε, και υψηλούς, υψηλότερου στόχου. Η Κομισιόν όμω πρέπει να εξισορροπήσει τι φιλοδοξίες με την ε, πραγματικότητα, με το ρεαλισμό. Και ελπίζω να το βλέπετε αυτό και να τενακλάτε αυτό στο κείμενο. Αυτό το κείμενο πιστεύουμε ότι μπορεί να σταθεί και μετά από μια μέθοδο ανάλυσης και να σταθεί σε μια κριτική δηλαδή. Ναι, θα πρέπει να ενδυναμωθεί το κείμενο αυτό σε διάφορα σημεία. Αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη δεσμευτούν, θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες εκθέσεις και λογοδοσία, θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο στεναροί ε, και αυστηροί απέναντι σε αυτούς που καθυστερούν, χρονοτριβούν και δεν προοδεύουν τα επόμενα χρόνια, αλλά επίσης θα πρέπει να δώσουμε και τα απαραίτητα κίνητρα από ευρωπαϊκής πλευράς, οικονομικά και άλλα, για να στηρίξουμε και τις προσπάθειες που κάνουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, περισσότεροι ή λιγότεροι στόχοι. Το βασικό θέμα είναι όχι να συμφωνήσουμε μόνο εδώ μεταξύ μας, αλλά και στο Συμβούλιο. Και για να υπάρξει συμφωνία πρέπει να υπάρχουν ε, στόχοι και πρέπει να υπάρχουν κρίσιμοι στόχοι, στόχοι κλειδιά για να βασιστεί η ευρύτερη ατζέντα, η οποία δεν αντιμετωπίζεται εξονυχιστικά στο κείμενο, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσετε ότι οι στόχοι που συμπεριλαμβάνονται είναι πιο κρίσιμοι, πιο βασικοί. Θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες, με ένα σχέδιο δράσης που θα αφορά συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε. Θα σας προτείνω μια ακόμα σειρά ερωτήσεων και αν κάποιοι συνάδελφοι ε, θέλουν να παρέμβουν θα κάνουμε ένα τελευταίο γύρο Catch the Eye. Αυτό το έγγραφο για τη στρατηγική 2020 που εγώ θα προτιμούσα να έχει ονομαστεί στρατηγική αλληλεγγύης και βιωσιμότητας φέρει το, τη σφραγίδα της δικής σας επιρροής, αλλά ε, φοβούμαι πως δεν θα ικανοποιήσει απόλυτα όλα τα μέλη της Επιτροπής, γιατί είδατε συμβαίνει αυτό με βάση τις παρεμβάσεις των συναδέλφων. Βέβαια, το έγγραφο αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενη διαβούλευση με του κοινωνικού εταίρου. Εγώ πάντω, αν ήμουν στη θέση σα, θα ήμουν σε δύσκολη θέση, γιατί ε, η θέση, η βάση μάλλον επί τη οποία έγινε η διαβούλευση ήταν ένα έγγραφο όπως θύμισε ο κύριος Σεμάν το οποίο εξεδόθηκε το 24 Νοεμβρίου 2009 ε, μια ημερομηνία που δεν ήσασταν εσείς ακόμα υπεύθυνο και όπου δεν φέρει ε, τη σφραγίδα των επιτρόπων που θα αναλάβουν να θέσουν σε εφαρμογή τη στρατηγική αυτή. Και αυτό για μας είναι ένα μήνυμα ότι η βάση επεξεργασίας αυτού του εγγράφου από την δημοκρατική άποψη ίσως να ε, δημιουργεί πρόβλημα. Και έπειτα βλέπω το, το χρονοδιάγραμμα όπως το προτείνατε στην τελευταία σελίδα του εγγράφου και με εκπλήσουν τα εξής. Καταρχήν, σε όλη την πρώτη φάση 2010 για την έγκριση του εγγράφου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αναφέρεται. Φαντάζομαι πως είναι ακόμα ένα σημάδι για την προνομιούχα συνεργασία με το Κοινοβούλιο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το εντάξει και το Κοινοβούλιο, γιατί αλλιώς θα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Και τα διαπιστώνουμε ότι τον Οκτώβριο εκ νέου προβλέπεται συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για θέματα επιλεγμένα και ίσως ήταν σκόπιμο να μας διευκρινίσετε κάπως ποια είναι το πνεύμα αυτής της διαβούλευσης. Ο κ. Κρίστενσεν μίλησε για το θέμα του κοινωνικού ντάμπινγκ και είπατε ότι δεν μπορούσαμε να προκαθορίσουμε το τέλος του κοινωνικού τάμπινγκ Ωστόσο, υπάρχουν εργαλεία για να αποφευχθεί το κοινωνικό τάμπινγκ και ανάμεσα σε αυτά υπήρχε ένα που είχαμε τη συνήθεια να το συζητάμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, γνωρίζω ότι δεν μπορείτε να βάλετε τα πάντα σε αυτό το έγγραφο που είναι περιορισμένο στη, ε, όσον αφορά τις σελίδες και τις σειρές. Το είπατε δύο φορές, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω γιατί μια λέξη μια ακροστοιχίδα με πέντε γράμματα δεν υπάρχει. Δηλαδή το ΣΣΣ τεμπέ. Δηλαδή η, βασι, η φορολογική βάση για τις ε, ε, επιχειρήσεις. Και όταν μιλάμε για κοινωνικό ντάμπινγκ και το θέμα της εναρμόνισης είναι ένα θέμα κρίσιμο. Ίσως όμως να μην διάβασα καλά το έγγραφο και κάπου να βρίσκεται αυτή η ακροστοιχίδα. Τώρα, κατά βάση εγώ θέλω να σας ρωτήσω και ένα συνάδελφο παρενέβη με, υπό το ίδιο πνεύμα πριν από λίγο και το είπατε και εσεί ο ίδιος, ότι τα δεκαετή προγράμματα είναι πολύ σημαντικά, αλλά δεν ξέρουμε πάντοτε τι θα συμβεί εντωμεταξύ. Και ίσω θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για τις ενδιάμεσες φάσεις. Και από αυτή την άποψη Πιστεύω πως είναι δύσκολο να μιλάμε σήμερα για την κατάσταση, για τη στρατηγική 2020, αν δεν δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γιατί τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή ζητά από τη χώρα αυτή να να αποδυναμώσει το κοινωνικό της πρότυπο ώστε μεθαύριο ο άρρωστος να πάει καλύτερα. Ενώ κατά τη διάρκεια όλη τη κρίση μας είπαν ότι το κοινωνικό πρότυπο το οποίο είναι ένας ε, αυτόματο σταθεροποιήτη είναι αυτός που είχε επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να περάσει ε, πιο εύκολα την κρίση από ότι αν δεν το είχαμε. Λοιπόν, πώς θα λυθεί αυτή η αντίφαση και μέσα στο ίδιο πνεύμα. Αν δούμε τον απολογισμό των όσων συνέβησαν μέσα στα χρόνια της στρατηγικής της Λισαβόνας βλέπουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Είχαμε τονίσει την ανάπτυξη και την απασχόληση, όμως σήμερα ο παράγοντας ανάπτυξη χρειάζεται ακόμα σε μεγάλο βαθμό γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξει ανάκαμψη και απασχόληση γιατί οι προοπτικές που έχουμε δεν ε, μας ικανοποιούν. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να πω στους πράσινους ούτε καν στους σοσιαλιστές ότι μιλάμε για ανάπτυξη έτσι γενικά και αόριστα. Θα πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, να είναι βιώσιμη. Γι' αυτό και λέω ότι αυτή η στρατηγική θα πρέπει να λέγεται στρατηγική αλληλεγγύης και βιωσιμότητα. Αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε πως αυτή η ανάπτυξη θα δημιουργήσει και θέσεις απασχόλησης. Γιατί στην προηγούμενη περίοδο μας εξήγησαν ότι πάνω από το 2% δεν χρειάζεται κανεί να ονειρεύεται να δημιουργεί θέσει απασχόληση. Τώρα οι προοπτικέ είναι κάτω από το 2%. Τώρα πρέπει να ξεπεράσουμε λοιπόν πρώτα το 2%. Αλλά εγώ αυτό που διαπίστωσα στην προηγούμενη περίοδο είναι ότι με ανάπτυξη πάνω από το 2% πολλέ φορέ δεν είχαμε και αντίστοιχη δημιουργία θέσεων. Πώ θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο και πώ, κύριε Επίτροπε, ίσω να χρησιμοποιήσουμε και το άρθρο 9, δηλαδή να υποχρεώσουμε του επενδυτέ να έχουν πραγματικέ στρατηγικέ όχι εγκατάσταση, αλλά απασχόληση μέσα στην Ένωση οργάνωση. Καταρχάς, ε, πιστεύουμε σοβαρά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό την επομένη ε, της δημοσίευσης του εγγράφου έρχομαι ενώπιόν σας να το συζητήσουμε και θα συνεχίσω να είμαι στη διάθεσή σας ε, όποτε χρειαστεί για οποιαδήποτε ε, μελλοντική συνεργασία. Από τη συνθήκη είμαστε υποχρεωμένοι να διαβουλευόμαστε για τις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση και αυτό θα γίνει άλλωστε και κατά τη διάρκεια της φετινής Άνοιξης και το είπα και στην εισαγωγική μου παρέμβαση. Διαβουλεύσεις έγιναν με τους κοινωνικούς εταίρους με βάση ένα άλλο κείμενο. Ε, προσωπικά ε, ε συνείδησαν ε, ηγέτες της Business Europe και των συνδικάτων για να συζητήσουμε, να ακούσω τις απόψεις τους εφόσον δεν συμμετείχα στη σύνταξη του ε, κειμένου και στην όλη διαδικασία πριν τα τέλη Ιανουαρίου. Από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι τούτη εδώ η νέα επιτροπή ε, είχε τελικά το τελευταίο λόγο. Διάφοροι επιτροπή συναρμόδιοι που ασχολούνται με τα σημαντικά θέματα, τις ναυαρχίδες και τους στόχους και έχουμε ε, σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην ολοκλήρωση και στην οριστικοποίηση του κειμένου. Είναι δικό μας δηλαδή το κείμενο της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, σύντομα θα έρθουν οι ενσωματωμένες ε, κατευθυντήριες γραμμές με μορφή δέσμης και στόχος είναι η συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην άλλη συζήτηση. Μερικά σημεία για την Ελλάδα. Βεβαίως ε, είναι αυτό κομβικό σημείο. Η αχίλιος πτέρνα θα έλεγε κανείς ε, της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας. Οι αδυναμίες οικονομικής και νομισματικής ένωσης έχουν καταδειχθεί τους τελευταίους μήνες. Και πάλι βέβαια η κατάσταση αυτή είναι κάτι που δεν βρίσκουμε στα περισσότερα εγχειρίδια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμετέχει οπωσδήποτε σε καμία περίπτωση με στόχο την υπονόμευση του κοινωνικού προτύπου. Συμμετέχουμε στη προσπάθεια σταθεροποίησης των δημοσίων οικονομικών της ΟΝΕ ναι, κατ' επέκταση, της Ευρωζώνης. Και στόχος είναι η δημιουργία διαφάνειας καθώς επίσης και ε, δημιουργία ισχυρών θεμελίων για βιωσιμότητα στα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε στο παρελθόν, σε προηγούμενες θέσεις απασχόλησης που είχα, είχα την ευκαιρία να μελετήσω και να συγκρίνω διάφορες ε, χρηματοπιστωτικές κρίσεις και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ελληνική περίπτωση δεν είναι η πρώτη περίπτωση χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε παρελθούσα εμπειρία και ε, στο συντονισμό των πολιτικών προσαρμογών ε, για να αποφύγουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με ε, την κυβέρνηση της χώρας ε, των κάστοτε κρατών μελών για να επιλέξουμε από την πιθανή έκβαση. Βέβαια, όταν επικρατεί τέτοιο πανικό στι χρηματαγορέ, είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει κανεί προ μια ιδεώδη λύση. Είναι ε, όμως σημαντικό να έχουμε επίγνωση και συνείδηση και της κοινωνικής διάστασης και της απασχόλησης. Και σε προηγούμενες περιπτώσεις ε, το γνωρίσαμε. Για να μην πάμε πολύ μακριά, στην Ουγγρική περίπτωση, όπου χρειάστηκε ακόμα πιο σκληρή δημοσιονομική προσαρμογή από τη, ε, τα γεγονότα αυτής της εβδομάδας. Αλλά κατάφερε η κυβέρνηση να ε, βρει μια λύση, ας πούμε, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και τους, ε, τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στη χώρα για να διασωθούν και να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και η απασχόληση. Υπάρχει λοιπόν εμπειρία που μπορούμε να μοιραστούμε τώρα, αλλά βεβαίως καταλαβαίνουμε την πάρα πολύ δύσκολη αφετηρία και για την ευρωπαϊκή οικονομία και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως χρειάζεται ανάπτυξη και θα πρέπει να τεθούν ξανά τα θεμέλια για την ανάπτυξη. Και ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί έχουμε ε, το εξής πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. πώς αντισταθμίζεται η μείωση του δυναμικού ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πώς θα αναζωογονηθεί για να υπάρχει μεγαλύτερη ανάπτυξη. Το ίδιο το δυναμικό. Δεν είναι εύκολο ερώτημα να απαντηθεί αυτό. Και η απάντηση που δίδεται είναι επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ενίσχυση της ανάπτυξης και ε, παιδείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ανάπτυξης, να δεσμευτούν περισσότερο τα κράτη-μέλη σε όλους αυτούς τους τομείς και έτσι βάσει των προσδοκιών μας θα έχουμε καλύτερο δυναμικό για ανάπτυξη. Αλλά δεν υπάρχει αυτοματισμός. Χρειάζεται πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κυβερνήσεων των κρατών μελών επίσης. On, uh, για το CCTV, για τη φορολογία. <laughs> Ξέρω ότι δεν είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, Άρα, ναι, ναι, ε, ήταν ε, θέμα του προηγούμενο επιτρόπου, Επιτρόπου και ευτυχώς έχω κληρονομήσει και ε, πολύ καλούς υπαλλήλους που μου βοηθούν πάρα πολύ από τον προηγούμενο επίτροπο και με βοηθούν για την φορολογική εναρμόνιση αλλά και πάλι το σημαντικό είναι και πάλι να αποφευθεί και το κοινωνικό dumping και το φορολογικό dumping και να ξεφορτωθούμε επιτέλους τις τρευλές ε, πρακτικές και είναι πολύ γνωστά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε ε, στην ιστορική αγορά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση αυτή. Βέβαια δεν είναι θέμα του χαρτοφυλακίου αλλά θα ξανάρθω να το συζητήσουμε. Euh, Διερωτώ με ποια ήταν η εντολή που δόθηκε στο Μάριο Μόντι μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Κύριε Σέρκα, θέλετε να παρέμβετε. Μία ερώτηση. Θα έχουμε καμία ευκαιρία να τροποποιήσουμε αυτό το έντυπο. Συγκεκριμένα ούτως ώστε να αντανακλώνται οι ανησυχίες μας. Ε, χαίρομαι που ο Επίτροπος αναφέρει κάποια στοιχεία της ε, κοινωνικής πολιτικής, αλλά δεν θέλουμε να είναι δευτερεύουσα σημασία σε αυτό το έγγραφο. Ας πούμε το θέμα της ε, μετανάστευσης που λέει το κείμενο. Θα έχουμε μια πλήρη πολιτική, ε, συνολική πολιτική για την πολιτική μετανάστευση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς αλλά δεν μιλάει καθόλου ας πούμε, για το ε, γραφείο, ε, Παγκόσμιο Γραφείο Εργασία. Δεν μιλάει καθόλου, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση για την ε, κοινωνική ένταξη. Πώς θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα. Πώς θα έχουμε την ευκαιρία ως Κοινοβούλιο να μιλήσουμε για αυτό το κείμενο. Ή δεν θα έχουμε την ευκαιρία. Κυρία Τσίμερ, μισό λεπτό. Και μετά τέλος. Τότε θα ήθελα να επανέλθω στο έγγραφο και να ρωτήσω το εξή συμπροματικά. Στη στρατηγική λέτε 20 εκατομμύρια μέχρι το έτος 2020 ε, που ζουν στο όριο της στόχιας, να μειωθεί αυτός ο αριθμός. Αυτό τι σημαίνει, ότι είστε πρόθυμοι να σκεφτείτε κάτι και να εφαρμόσετε όμως συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μειωθεί Αυτό, δηλαδή το, το όριο της στόχης που είναι το 60% για τα νοικοκυριά του ε, εθνικού ΕΠ, θα το συζητήσετε αυτό με τα κρατημέλη, θα το εφαρμόσετε με τα κρατημέλη μαζί. Εγώ είμαι πρόθυμος πάντα να συζητώ όλα αυτά τα θέματα ε, σε όλη την ε, για όλη την Ευρώπη στις προδιαγραφές βέβαια. Υπάρχει μια ιδέα που τη λέει ήδη το έγγραφο ε, που λέει ότι θα πρέπει κάθε φορά να υπάρχουν προγράμματα αναπερίπτωση, κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του κράτους μέλους. Ε, είναι άνισα μεταξύ τους τα κράτη-μέλη, δεν έχουν ίδιες συνθήκες, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα μοντέλο σε μία χώρα και να την εξάγουμε σε μία άλλη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα υποστηρίζει το εκάστοτε κράτος μέλος να αναπτύσσει τις δικές του μεθόδους για να περιορίζει τη φτώχεια. Οι δείκτες της φτώχειας και τα ποσοστά της φτώχειας ερμηνεύονται στο εσωτερικό μιας χώρας και τελικά θρίζονται για να φτάσουν στους αριθμούς που λέμε στο έγγραφο. Αλλά είναι ένα θέμα της κάθε χώρας και ο στόχος είναι εφικτός. Ε, όταν συμφωνούμε και πηγαίνουμε προς την ίδια κατεύθυνση, γιατί να αλλάξουμε το κείμενο όταν έχουμε την ίδια ε, αντίληψη και τα ίδια αιτήματα. Σήμερα άκουσα ε, από τη μια ε, λέτε ότι δεν είναι αρκετά φιλόδοξο, άλλοι λένε ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο και είναι πολύ σκεπτικιστές ως προς τους στόχους, ιδιαίτερα το στόχο της φτώχειας. Ε, τώρα τι να σας πω. Εμείς ακούμε, συζητούμε και ελπίζω τα συμπεράσματα να είναι τα ορθά. Αλλά ο διάλογος με το Κοινοβούλιο θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όπως βλέπετε όταν σε εγκρίνει μετά από κρόαση το Κοινοβούλιο σε Επίτροπο, μετά από απαιτητική ακρόαση, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο εύκολες οι συζητήσεις μετά. Τα μέλη μας είναι απαιτητικά, αλλά αυτό είναι ο ρόλος των βουλευτών. Να ε, φέρνουν ενώπιον των ευθυνών στην εκτελεστική εξουσία. Πήρατε μια πρώτη γεύση σήμερα. Ε, Έπετε και συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε ένα διάλογο έτσι, με εμπιστοσύνη. Τελειώσαμε εδώ τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ραντεβού την επόμενη φορά στις 16 και 17 του μηνός.